Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, αρχίζουμε τη συνεδρίασή μας για σήμερα το απόγευμα. Έχουμε δημόσια ακρόαση. Έχετε την ημερήσια διάταξη. Θα συζητήσουμε για τις επιστημονικές και πανεπιστημιακές σταδιοδρομίες και για τους αόρατους φραγμούς. 24 Νοεμβρίου 2014 έδωσε το Προεδρείο την άδειά του για ακρόση της Επιτροπής μας στα πλαίσια του πρώτου εξαμήνου του 2015. Έχουμε τέσσερις εμπειρογνώμονες εδώ μαζί μας που θα πάρουν και το λόγο με τη σειρά. Πρώτα απ' όλα να σας ε, παρουσιάσω την κυρία Μελίσα Ρανκούρου, η οποία είναι από την ε, μη κυβερνητική οργάνωση Πράσινο Φως για τα Κορίτσια από το Βέλγιο. Στη συνέχεια θα ακούσουμε την κυρία Μεριάννα Νέντοβιτς, η οποία είναι από την Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών Λάβος Λάβα Ρούτσισκα στο Βούκοβαρ της Κροατίας. Καλώς ήρθατε. Στη συνέχεια θα δώσω το λόγο στην κυρία Στρέλα Μόντες Λόπες, που είναι από το Τμήμα Κοινωνιολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου του Σαλαμάνκα στην Ισπανία. Και τέλος, ο τελευταίος προσκεκλημένος μας είναι ο κύριος Πέτερ Ντρέλ, που είναι ε, διευθυντής της, ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Διεύθυνσης για την Καινοτομία και την Έρευνα. Καλώς ήρθατε όλοι. Η ακρόαση αυτή πιστεύω θα μας δώσει πολλές επιπλέον πληροφορίες όσον αφορά την έκθεση πρωτοβουλίας που φέρει τον ίδιο τίτλο. Η εισηγήτρια δυστυχώ δεν θα είναι εδώ. Έχουμε όμως την κυρία Λεγκρίπ που παίρνει τη θέση της. Στην συνεδρίαση μας του Ιουνίου θα εξετάσουμε για πρώτη φορά την έκθεση αυτή. Λοιπόν, θα δώσω το λόγο πρώτα στην κυρία Ρανκούρ. Thank you. Σας ευχαριστώ. Είναι τιμή μου να μιλήσω για το θέμα. Αγαπώ τις επιστήμες. Την κάθε τους πτυχή. Την ανακάλυψη, το πείραμα, τις καινοτομίες τους. Είναι υπέροχο αντικείμενο και αφορά όλη μου τη ζωή. Από πολύ νεαρή ηλικία ήξερα ότι οι επιστήμες και όλα τα σχετικά ε, αντικείμενα, τα μαθηματικά, η πολιτική μηχανική, αυτά που σήμερα ονομάζονται θετικέ επιστήμε, θα ήταν ένα ενεργό μέρο τη ζωή μου. Αφού διάβασα ένα βιβλίο για τι γυναίκε στο Πολυτεχνείο από την δόκτωρα Λίλιαν Γκίλπερ, όταν ήμουν μόλι 12, Πραγματικά ε, μου φάνηκε συνεργαστική ιδέα να γίνω πολιτικό μηχανικό. Και με ενθάρρυνε και η μητέρα μου να φτάσω το όνειρο αυτό. Ε, με το όνειρο αυτό λοιπόν το πέτυχα και κατάλαβα να έχω την πρώτη, κατάφερα να έχω την πρώτη μου δουλειά στα 19. Έτσι ξεκίνησε μια σταδιοδρομία που πάντοτε συμπεριλάμβανε τις επιστήμες, την πολιτική μηχανική και τα μαθηματικά. Όμως ε, σε όλες τις καλές ιστορίες και σε κάθε ταξίδι υπάρχουν και τριγμοί που ε, φαίνονται σαν εμπόδια μέχρι να φτάσει κανείς στο στόχο του. Εμένα τα εμπόδια αυτά συμπεριλάμβαναν το να μου λένε οι καθηγητές και άλλοι ότι δεν ήμουν αρκετά καλή και να το πιστεύω. Ε, και υπήρχε αρνητικό, ε, αρνητική διάθεση στις ε, πανεπιστημιακές ομάδες για τις γυναίκες. Υπήρχαν διαρκώς απορίες και ερωτήσεις για την ανάγκη να συμμετέχει μια γυναίκα σε ομάδα πολιτικών μηχανικών και το ίδιο με γραφίτι που πολλές φορές σε τείχους ζωγραφίζονταν με συνθήματα κατά των γυναικών στις πολυτεχνικές σχολές. Με έχουν πει και ακόμη και αν ήταν βρισιά θα ήταν ε, περίεργο. Επίσης ο μόνος λόγος που μου είπαν ότι βρήκα δουλειά είναι επειδή είμαι γυναίκα. Αυτή και ήταν και η πρώτη μου θέση και ήμουν τόσο ενθουσιασμένη όταν ξεκινούσα. Όμως ξαναπήγα στην ομάδα μηχανικών ε, όλους, ε, όλοι οι άντρες με τους οποίους ήμουν στο πανεπιστήμιο τους είπα βρήκα την πρώτη μου δουλειά και μου είπανε μπράβο σου επειδή είσαι γυναίκα μάλλον θα τη βρήκες και όχι και πριν από τόσο καιρό, πριν από καμιά διετία περίπου, είχα μια καταπληκτική ευκαιρία επαγγελματική με μια συνέντευξη εργασίας λίγα λεπτά από το σήμα που βρισκόμαστε σήμερα και μιλούσα για την καριέρα του συζύγου μου στην ε, συνέντευξη αυτή και τα σχέδια που είχα για να αποκτήσω παιδιά. Αυτά με ρωτάγανε και ήταν και μια διεθνή οργάνωση επιστημών. Εγώ ήμουν από τι τυχερέ παρόλα αυτά. Αυτό είναι μόνο κάποιε από τι ιστορίε που μπορεί να ακούσει κανεί και σίγουρα δεν θα είχα βρει το δρόμο μου ε, και δεν με εμπόδισε να πετύχω του στόχου μου αυτή η νοοτροπία. Αλλά Όλα αυτά δεν με εμπόδισαν σε κανένα βαθμό. Απλώς με ανάγκασαν να σκεφτώ και να σκεφτώ ξανά πώς θα πρέπει να μείνομαι, πώς θα οργανώσω το μέλλον μου και μου έδωσαν και τα κίνητρα για να συνεχίσω και να επιδιώξω με ενθουσιασμό το σκοπό μου. Η ιστορία, η προσωπική, η δική μου, είναι ένα μικρό παράδειγμα που το δείχνουν και οι στατιστικές, δείχνουν τη σκληρή πραγματικότητα σήμερα. Οι αριθμοί, οι έρευνες και οι μελέτες θα σας πούν ότι οι σταδιοδρομίες, η ακαδημαϊκή καριέρα και οι σπουδές ε, στα πολυτεχνία είναι εξαίρεση για τις γυναίκες. Στις θεστικές μας δείχνουμε, βλέπουμε ότι η αυτοεκτίμηση των γυναικών ε, πέφτει σε μια συγκεκριμένη ηλικία, γύρω στα 11. Το επίπεδο αυτοεκτίμηση εκεί είναι γύρω στα 70 και όταν φτάσουν ε, στα 15 το ποσοστό της αυτοπεποίθησης πέφτει στα 55%. Το 1 πέμπτο των ε, γυναικών που φοιτούν σε πολυτεχνικές σχολές ε, αναρωτιούνται αν ανήκουν εκεί. Μόνο το 20% των ε, γυναικών με πτυχία σε τέτοιους τομείς έχουν ανάλογη θέση εργασίας και είναι πολύ μικρό το ποσοστό των γυναικών που είναι φοιτήτριε σε τάξεις και αμφιθέατρα με πολιτικούς μηχανικούς και είναι ακόμα λιγότεροι αυτοί που τελικά μένουν σε αυτή τη δουλειά. Ε, υπάρχουν οργανισμοί που λένε ότι Υπάρχουν πολύ λίγες γυναίκες μηχανικοί ε, στην ομάδα που εκπροσωπείται από αυτή τη διεθνή οργάνωση. Μόνο 10% των κοριτσιών μάλιστα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούν ότι ε, μπορούν να κάνουν επιστημονική καριέρα. Ένα στα τρία κορίτσια παντρεύεται πριν τα 18 και οι περισσότερες εγκαταλείπουν το σχολείο πριν καν παντρευτούν. Όλα αυτά συμβαίνουν διότι Υπάρχει ακόμα προκατάληψη και γι' αυτό συμμετείχα σε μια κερδοσκοπική οργάνωση πριν από λίγα χρόνια για να καταπολεμηθούν οι προκατάληψει κατά των γυναικών. Ε, τα τελευταία χρόνια ε, έχουν ε, στατολογηθεί τουλάχιστον 1.500 εθελοντέ από τέτοιε οργανώσει και μιλήσαμε με χιλιάδε παιδιά σε πέντε υπήρου και θέλαμε να του δείξουμε ότι είναι και διασκεδαστικέ και απαραίτητε οι επιστημονικέ σπουδέ. Το αποτέλεσμα είναι ότι 94% των παιδιών που συμμετείχαν σε αυτό το πρόγραμμα τελικά θα αρχίσουν να σπουδάζουν θετικέ επιστήμε και δεν ξέρουμε αν θα είναι μόνο καθοριστική διαφορά, αλλά είναι πιο ενδιαφέρον ότι οι νεαροί αυτοί άνθρωποι μπορεί να πετύχουν κάτι και οι γονείς τους είναι υπερήφανοι που θα ακολουθήσουν τα όνειρά τους. Οι ιστορίε αυτών των παιδιών είναι πολύ ε, ενδιαφέρουσε. Η Τζάκη δημιούργησε μια εφαρμογή στην ηλικία των 12. 12. Η Σάρα δεν γίνεται δεκτή σε μια ε, ομάδα νεαρών επιστημόνων. Η Σεσίλια ήδη ξεκινήσει τι σπουδέ και σκέφτεται να πάει στο Πανεπιστήμιο στο Πολυτεχνείο αλλά και οι γονείς. Οι γονείς μας ευχαριστούν που φέραμε τις επιστήμες στη ζωή των παιδιών τους. Ε, οι ελπίδες μας για το μέλλον είναι ότι οι γυναίκες δεν θα αποθαρρύνονται από οποιοδήποτε όριο μπορεί να τους επιβληθεί και ότι ε, η ελπίδα αυτή γιατί θα συνοδεύσει την πολλή δουλειά που πρέπει να κάνουμε. Οι γυναίκες στις επιστήμες και στα πολυτεχνία ε, πρέπει με πρωταγωνιστικό ρόλο να προβάλλουν ε, την περαιτέρω δράση που χρειάζεται και να αντιμετωπιστούν οι φραγμοί που σήμερα οι γυναίκες ε, επιβάλλονται στις γυναίκες, στις επιστήμες και σε άλλους τομείς. Ένα μικρό, μια μικρή γεύση είναι αυτή για το πώς είναι να είναι κανείς δεκάχρονο σήμερα. Δείτε αυτό το κλιπ και θα καταλάβετε καλύτερα.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

Αυτή είναι μια πρώτη ιδέα. Έχει να κάνει με την αυτοπεποίθηση και τις στατιστικές που σας ανέφερα. Δηλαδή ένα 10χρονο, 11χρονο κορίτσι ε, στο επίπεδο της αυτοπεποίθησης φτάνει το 75% και λίγα χρόνια μετά. Αυτό το ποσοστό φτάνει το 55% και αυτό συνεχίζεται. Πραγματικά διστάζω ε, να ρωτήσω τι θα συνέβαινε με κάθε μια από εμά αν να μα ρωτούσαν. Η πρώτη ιδέα, η πρώτη δράση θα ήταν η αυτοπεποίθηση των 10 χρόνων να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα. Ένα τρόπο να γίνει αυτό είναι να κοιτάξουμε οι οργανώσεις πώς μπορούν να ενθαρρύνουν τις θετικές σπουδές. Πρέπει οι γυναίκες να ενθαρρύνονται, να σπουδάζουν ε, τα προγράμματα των θετικών επιστημών. Ίσως ξεκινώντας από το γυμνάσιο, το λύκειο, το πανεπιστήμιο θα πρέπει να μπορούν οι μαθητές και φοιτητές να δουν πού μπορεί να είναι το μέλλον τους. Και ε, επιμένω σε αυτό, γυμνάσιο, λύκειο και πανεπιστήμιο. Αυτή την ηλικία στοχεύουμε. Τότε είναι τα παιδιά που ψάχνουν και αναρωτιούνται για τις δουλειές τους. Περισσότερος ανταγωνισμός ε, για την καινοτομία των ε, επιστημών σε όλα τα επίπεδα. Οι εταιρείε όπω η Cisco δημιούργησαν ε, πολλέ νέε ιδέε να ενθαρρύνουν παιδιά να βρουν καινοτομίε που μπορούμε να τι χρησιμοποιήσουμε σήμερα στην κοινωνία μα και να γίνουν διατρατικέ επιστήμε, ε, χρήσιμε και με νόημα σε όλα τα επίπεδα τη ε, παιδεία. Για να μπορεί η εκπαίδευση και το εκπαιδευτικό σύστημα να κάνει τα παιδιά να συμμετέχουν και να έχουν ενδιαφέρον για αυτέ τι σπουδέ. Α κοιτάξουμε λοιπόν γιατί η αυτοπεποίθηση ενό δεκάχρονου μπορεί να μειώνεται καθώ μεγαλώνει. Α σπάσουμε του φραγμού που πρέπει να αντιμετωπίσει αυτό το δεκάχρονο και να προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε τη συμμετοχή τη στο επιστημονικό πεδίο. Να τη δείξουμε ότι τα πάντα είναι δυνατά. Αυτό θα έλεγα σήμερα στα νερά κορίτσια και ότι είναι εφικτό. Το δεύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι κάτι που αφορά εμάς προσωπικά, δηλαδή οι δράσει ε, που, κάνουμε εμείς, που αναλαμβάνουμε εμείς οι ίδιοι και που αφορούν εμάς εδώ. Ε, δηλαδή, να ενθαρρύνουμε κάποιον γνωστό μα, τον δικό μα τον κύκλο, να κάνει το ίδιο. Α αναλάβουμε λοιπόν τη δράση, να βελτιώσουμε τι δεξιότητέ μα και να μην αφήσουμε κανένα φραγμό, κανένα εμπόδιο να μπει μπροστά στα όνειρά μα και στου στόχου μα. Πώ μπορεί να γίνει αυτό, Μπορούμε όλοι να δημιουργήσουμε ένα επαγγελματικό δίκτυο εντό ή εκτό τη εταιρεία μα, τη περιφέρειέ μα ή του τομέα μα. Μπορούμε να λειτουργήσουμε ως μοντέλα και πρότυπα και ως μέντορες και να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τις δεξιότητές μας με νέα θέματα, με, νέες, ε, με νέους τομείς, με νέες διδασκαλίες. Ε, θα πρέπει να μην χάνουμε καμία ευκαιρία και να σκεφτόμαστε ότι δεν πρέπει να λέμε ναι αυτόματα, αλλά να σκεφτόμαστε και το ναι. Ε, θα πρέπει λοιπόν κάθε ευκαιρία να την αρπάζουμε, να την μελετούμε και αυτό το έκανα εγώ σε κάθε περίπτωση, ασχέτως με το τι είχα να αντιμετωπίσω. Και τέλος, αυτό που μπορούμε όλοι να κάνουμε για να υπάρχει και ε, κάποιο είδου εσωτερική γνώση για τους υπόλοιπους οργανισμούς, είναι να τις ενθαρρύνουμε, να προβλέψουν ευφιέστερα συστήματα για να μπορέσουν οι γυναίκες να αναλάβουν ενεργό ρόλο στις επιστήμες και να έχουν και πρωταγωνιστικούς ρόλους. Δηλαδή δεξιότητες, ίσες ευκαιρίες και ε, ίση μεταχείριση. Να δημιουργηθούν άτυπα και επίσημα δίκτυα στις εταιρείε με μισθολογική αναθεώρηση βάσει των, ε, της εγκριτικής αξιολόγησης της αγοράς που να λαμβάνουν υπόψη την ισότητα των φύλων με πολιτικές που να θαρρύνουν τόσο τις μητέρες όσο και τους πατέρες να βοηθούν τα παιδιά και με εκπαιδευτικέ ευκαιρίες που να οδηγούν στη δημιουργία πρωταγωνιστών. Το όνειρό είναι απλό. Μια μέρα μία γυναίκα από τις επιστήμες του Πολυτεχνείου ή οποιαδήποτε άλλη καριέρα θα αναλάβει μια γυναικα απο τι επιστημε του πολυτεχνειου η οποιαδηποτε αλλη καριερα θα αναλαβει μια δουλεια και χωρί ε, ε, καμία, ε, κανένα δισταγμό θα έχει την αυτοπεποίθηση ότι την πήραν όχι γιατί είναι γυναίκα αλλά γιατί μπορεί να συνεισφέρει τα μάλλα στην εταιρεία και να προσφέρει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, τον ηγετικό ρόλο που χρειάζεται αυτή η κοινωνία. Ήρθε λοιπόν η στιγμή να σπάσουμε τη γυάλινη οροφή και να την κομματιάσουμε κιόλα. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Το όνειρό σας είναι και το δικό μας όνειρο και γι' αυτό συζητάμε τα θέματα αυτά εδώ. Πρωτού δώσω το λόγο στο δεύτερο μιλητή. Θα ήθελα να καλωσορίσω τους οκτώ ε, προσκεκλημένους από το Ινστιτούτο της Νοτιής Κορέας για την ισότητα μεταξύ των φίλων. Σας καλωσορίζουμε. Θα δώσω το λόγο τώρα στην κυρία Μιλιάνα Νέντοβιτς από την Κροατία. Εκτός μικροφώνου. Eh, odnosno eh, tema je stakleni strop položaj žena u sustavu znanosti. Stakleni strop je pojam koji se koristi... Θα σας μιλήσω για αυτούς τους αόρατους φραγμούς. Την κρυστάλλινη οροφή, όπως τη λέμε, είναι μια έκφραση που δηλώνει ότι μία γυναίκα δεν μπορεί να προχωρήσει στη σταθεροδρομία της. Η θέση της γυναίκας αλλάζει σήμερα. Οι γυναίκες είναι πιο μορφωμένες και θέλουν, επιθυμούν να παίρνουν θέσεις πιο ψηλά στην ιεραρχία. Όμως η πιο καλά πληρωμένη δουλειά δίνεται στους άντρες και ακόμα και αν οι γυναίκες ανοιχτά ε, το λένε, ε, ποιες είναι οι φιλοδοξίες τους και ποιες είναι οι γνώσεις τους, δεν τα καταφέρνουν. Η θέση που κατέχουν πάντως στην εργασία είναι όλο και πιο σημαντικές. Έχω κάνει μια έρευνα και τα συμπεράσματα μας δείχνουν πού βρίσκεται η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην εργασία. Θα μπορούσαμε στην πραγματικότητα να μιλήσουμε πιο πολύ για ανισότητα στην εργασία και όχι για ισότητα στον τομέα των επιστημών. Στην Κροατία η κατάσταση δεν είναι αρκετά καλή. Ακόμα και αν οι γυναίκες μέχρι την ηλικία των 50 ε, προχωρούν στις σπουδές πιο πολύ από ότι άντρες, δεν κατέχουν αντίστοιχες θέσεις στην εργασία. Οι ηγετικέ θέσεις συνήθως δίνονται στους άντρες και δεν υπάρχουν αρκετά περιθώρια για τις γυναίκες. Ο όρος αυτός λοιπόν του κρυστάλλινου, της κρυστάλλινης οροφής είναι ένας όρος και ο άλλος όρος είναι ο λαβύρινθος. Είναι πιο σύγχρονη ορολογία αυτή, είναι μια μεταφορά που δηλώνει ότι ορισμένες γυναίκες καταφέρνουν να έχουν καλή δουλειά, δεν καταφέρνουν όμως να την κρατήσουν αυτή την καλή δουλειά. Γι' αυτό και πρέπει να μιλάμε για, αυτά τα, για αυτούς τους αόρατους φραγμούς. Αναρωτιόμαστε πώς θα λυθεί αυτή η κατάσταση. Το Πανεπιστήμιο του Ρίξ στην Κροατία 40 χρόνια είχε μία πρίτανη. Κάτι το οποίο δείχνει ότι στον κόσμο των γυναικών οι ηγετικές θέσεις καλύπτονται από τους άντρες. Δεν υπάρχει διάκριση, λένε ορισμένη βάση του φύλου. Τα δεδομένα όμως δείχνουν ακριβώς το αντίθετο. Στην Κροατία υπήρξαν αλλαγές όσον αφορά ηγετικές θέσεις που κατέχουν οι γυναίκες. Οι αλλαγές όμως είναι πραγματικά ελάχιστες, απειροελάχιστες. Οι στατιστικές δείχνουν ότι στον κόσμο των επιστημών υπάρχουν ακόμα σήμερα λόμπι αντρών, τα οποία εμποδίζουν τις γυναίκες να προχωρήσουν. Οι επιστημονικές πρόοδοι στην Κροατία περιλαμβάνουν 10 20% γυναίκες. Κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, είναι ιδιαίτερα απογοητευτικό. Οι γυναίκες όμως προσπαθούν να ξεπεράσουν τα εμπόδια. Πώς να σπάσουμε αυτόν τον όρητο φραγμό. Πρέπει να ρωτηθούμε τα εξή. Πρώτα απ' όλα, γιατί όταν έχουν ίδια προσόντα τελικά προσλαμβάνονται λιγότερες γυναίκες σε ηγετικές θέσεις. Δεύτερον, γιατί οι γυναίκες ακόμα και αν ε, στα πανεπιστήμια είναι περισσότερες, στις ηγετικές θέσεις είναι λιγότερες από ότι άντρες. Ποιοι είναι αυτοί οι αόρατοι φραγμοί. Η γυναίκα πάβει να είναι μια καλή γυναίκα, η μητέρα, σύζυγος, η μητέρα, αν ακολουθεί διοδρομία; Αν παρακολουθήσουμε την κατάσταση που επικρατεί στα πανεπιστήμια, Τη χρονιά 2013 με 2014, 28,6% των γυναικών γράφτηκαν. Δίπλωμα το 2013, το 58% ήταν γυναίκες. Η κατάσταση είναι η ίδια και για αυτούς που παίρνουν ε, μάστερ ή διδακτορικό. 57% παίρνουν μάστερ, κάνουν ειδικέ σπουδέ δηλαδή και 54% είναι αυτές που πήραν διδακτορικό. 57% είναι γυναίκες δηλαδή από αυτές που παίρνουν διδακτορικό. Κάτι το οποίο δείχνει ότι όταν μιλάμε για αυτό το κρυστάλλινο ταβάνι, αυτή την οροφή, τη γυάλινη, αυτή η μεταφορά συμπεριλαμβάνει όλα τα εμπόδια, τα όρατα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στη δουλειά τους. Ασχολήθηκα με αυτή την κατάσταση όσον αφορά τα επιστημονικά τμήματα στο Στρόσμαγερ Πανεπιστήμιο του ΟΣΕΓΕΚ. Κατάφερα λοιπόν εκεί να αναλύσω την κατάσταση και να δω πόσες θέσεις ηγετικές κατέχονται από γυναίκες σε 11 σχολές στο Πανεπιστήμιο αυτό του ΟΣΕΓΕΚ. Το συμπέρασμα είναι ότι είναι πολύ λίγες οι γυναίκες ή που εκπροσωπούνται στο Πανεπιστήμιο αυτό όσον αφορά τις ηγετικές θέσεις. Ε, από τις 11 σχολές, 10 σχολές έχουν Πριτάνης άντρες. Μόνο μία σχολή, μόνο εκείνη της φιλολογίας, έχουν γυναίκα πρίτανη. Αυτά είναι στατιστικά δεδομένα που μιλάνε από μόνα τους βέβαια. Αυτή είναι μια κατάσταση δύσκολη για τις γυναίκες όταν μιλάμε για την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Τώρα, η κατάσταση όσον αφορά τους αντιπρίτανες είναι λίγο καλύτερη. 42% των αντιπριτάνιων είναι γυναίκες. Και 58% είναι άντρες. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι γυναίκες έχουν περισσότερες δυσκολίες για να καταφέρουν να προχωρήσουν στη σταδιοδρομία τους και να καταλάβουν ηγετικές θέσεις. Πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχει ανισότητα τελικά μεταξύ ανδρών και γυναικών. Τέλος, αυτό που θέλω να προσθέσω είναι ότι αυτά τα, αυτή η αόρατη φραγμή είναι πραγματική. Μπορούμε να μιλήσουμε και για τον λαβύρινθο. Εγώ αναφέρομαι κυρίως στο τι συμβαίνει με τις επιστημονικές σταδιοδρομίες. Κανονικά θα πρέπει να είχαν τις ίδιες δυνατότητες οι άντρες και οι γυναίκες να ισχύουν ακριβώς τα ίδια και να έχουν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα. Το 2008 εγκρίθηκε νομοθεσία για την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Για την περίοδο 2011 με 2015 ακολουθήθηκε μια στρατηγική για την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Οι νομοθετικές πράξεις όμως δεν πρόκειται να αλλάξουν τίποτα αν δεν εφαρμόζονται κιόλα. Δεν φτάνει να περάσει ένας νόμος. Πρέπει να φροντίζουμε για την εφαρμογή τους όλα δείχνουν ότι στον κλάδο των επιστημών στην Κροατία υπάρχει ανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Πρέπει να φροντίσουμε να σπάσουν επιτέλους αυτά, αυτή η αόρατη φραγμή που υπάρχουν. Οι άντρες δεν θα το κάνουν από μόνοι τους. Οι γυναίκες πρέπει να φροντίσουν για την αλλαγή. Οι γυναίκες πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι είναι θύματα διάκρισης και να διταθούν. Ευχαριστώ πολύ. Ehm, Σα ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση αυτή. Πρόκειται για μια ακρόαση και ως εκ τούτου υπάρχουν λοιπόν ε, δυνατότητες ε, να θέσουμε και ερωτήσει προς τους αξιότιμους προσκεκλημένους μας. Καταρχάς όμως θα ήθελα να δώσουμε τη δυνατότητα να πάρουν το λόγο οι ομιλητές μας. Η κυρία Στρέγια Μόντες Λόπες έχει τώρα το λόγο. Παρά την πρόοδο που έχουμε σε θέματα ισότητας και τα βλέπουμε στα πανεπιστήμια τα τελευταία χρόνια, παρόλα αυτά η γυναίκα δεν μπορούμε να πούμε ότι βρίσκεται ακριβώς στην ίδια θέση με τους άντρες σε ηγετικές θέσεις, σε θέσεις μεγαλύτερου κύρου, εξουσίας και καλύτερων αμοιβών. Εδώ μιλάω για την ακαδημαϊκή βέβαια σταδιοδρομία, αλλά μιλάω επίσης και για την ε, πρόσβασή τους ως επικεφαλής τμήματων σε διάφορες σχολές στα πανεπιστήμια. Όσον αφορά τώρα τις διοικητικές θέσεις, συνήθως είναι κάτι που ξεχνάμε στις ερευνές μας όταν κάνουμε ερευνές στα πανεπιστήμια. Δεν έχω χρόνο βέβαια να πω λεπτομέρειες, αλλά το αναφέρω παρόλα αυτά. Στις διάφορες έρευνες που έχουν γίνει τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και πιο συγκεκριμένα σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, προσπαθεί να γίνει συνδυτοποίηση και να καταλάβουν ποια είναι η δυναμική που υπάρχει στα πανεπιστήμια και που εμποδίζει την πρόθεση των γυναικών και δεν τους δίνει τις ίδιες ευκαιρίες για να φτάσουν σε ηγετικές θέσεις. Το θέμα του φίλου είναι πολυεπίπεδο. Οι ίδιοι ακαδημαϊκοί δίνουν διάφορες εξηγήσει, εξηγούν σε διαφορετικά επίπεδα την κατάσταση. Στην πραγματικότητα όμως έχουν άμεση σχέση μεταξύ τους. Εγώ χρησιμοποιώ στην δικιά μου την έρευνα το θεωρητικό πλαίσιο μιας Ιρλανδικής έρευνας που έχει γίνει και θα σας αναπτύξω τις πιο σημαντικές έννοιες της έρευνας αυτής και θα σας δώσω στη συνέχεια πιο συγκεκριμένα παραδείγματα από την Ισπανία. Τα επίπεδα στα οποία αναφέρομαι είναι το ατομικό επίπεδο, το οργανωτικό επίπεδο δεύτερον και τρίτον το θεσμικό επίπεδο. Στο ατομικό επίπεδο ε, ακούμε διάφορες εξηγήσεις που λένε ότι φταίει η ίδια η γυναίκα. Δηλαδή ότι η γυναίκα είναι εκείνη η οποία έχει φτάσει σε αυτήν την κατάσταση, κάτι όμως που την επηρεάζει ψυχολογικά και δημιουργεί φραγμούς που το ακούσαμε και πριν δεν έχει αρκετή εκτίμηση στον εαυτό της, νιώθει ενοχές, ανασφάλεια κλπ. κλπ. Όλα αυτά οδηγούν η ίδια γυναίκα να αποφασίζει να μην συμμετέχει σε διαγωνισμούς, να μην είναι υποψήφια σε ηγετικέ θέσεις και να μην υποστηρίζει τα δικαιώματά της. Ενώ οι άντρες το κάνουν όταν, για παράδειγμα, προσπαθούν να πετύχουν καλύτερα ωράρια. Αυτό σημαίνει ότι οι άντρες και οι γυναίκες στα πανεπιστήμια πολλές φορές εξηγούν την δυσκολία αυτή η πρόσβαση σε ηγετικές θέσεις των γυναικών με το ότι η γυναίκα είναι αυτή η οποία αποφάσισε να μην συμμετάσχει στους σχετικούς διαγωνισμούς, να μην είναι υποψήφια. Η γυναίκα μπορεί να το αποφασίζει, αλλά στην πραγματικότητα η απόφαση της αυτή εξαρτάται από διάφορους παράγοντες που έχουν να κάνουν με την οικογενειακή της ζωή, για παράδειγμα. Αυτό το επιχείρημα πάντως, το ότι η γυναίκα φταίει, είναι αρκετά ελκυστικό. Όταν ε, αποφασίσουμε ότι η γυναίκα φταίει, ε, δεν θα κάνουμε απολύτως τίποτα, δεν θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τίποτα για να βοηθήσουμε τις γυναίκες. Δεύτερον, σε επίπεδο οργανωτικό. Τι λένε οι ίδιοι ακαδημαϊκοί αναφέρονται στην επίσημη δομή της οργάνωσης, αλλά και στην ανεπίσημη, δηλαδή στην οτροπία την οργανωτική που ισχύει. Και λένε, και μάλλον αυτά όμως δείχνουν ε, ότι τελικά το πανεπιστήμιο και η οργάνωσή του δεν είναι ουδέτερη απέναντι στα φύλλα. Στην ακαδημαϊκή σταδιοδρομία πρέπει να πούμε ότι αυτή οργανώνεται από εκείνους οι οποίοι φτάνουν στις ηγετικές θέσεις. Και ποιοι είναι αυτοί, οι άντρες βέβαια. Η ακαδημαϊκή σταδιοδρομία σχεδιάζεται από άντρε για άντρε. Στην έρευνα λοιπόν που έχω κάνει εγώ στην Ισπανία δείχνει ότι οι άντρε και οι γυναίκε τη σταδιοδρομία στην Ισπανία την βλέπουν σαν μια σταδιοδρομία ουσία που δεν μπορεί κανεί να διακόψει, ούτε ε, μπορεί να πει όχι αν χρειάζεται να δώσει χρόνο από την ιδιωτική του ζωή. Πρέπει να είναι διαθέσιμο μέρα, νύχτα να μπορεί να κάνει έρευνα ανα πάσα στιγμή. Μόνο έτσι μπορεί να προχωρήσει τη σταδιοδρομία του ερευνητή. Εφόσον λοιπόν πρόκειται για μια σταδιοδρομία που δεν μπορεί κανείς να διακόψει, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για μια γυναίκα η οποία θα φέρει στον κόσμο το παιδί της. Αν πρέπει να χρησιμοποιεί κανείς τον χρόνο του από την ιδιωτική του ζωή για να προχωρήσει στη αυτονομία ερευνητική, καταλαβαίνετε ότι αμέσως δημιουργείται ανισότητα μεταξύ αντρών και γυναικών, γιατί στην κοινωνία είναι διαφορετική η ρόλη της γυναίκας και του άντρε. Οι άντρες δεν συμμετέχουν εξίσου στην οικογενειακή ζωή, στην παιδική μέρημνα. Επιμένω στο ότι εδώ δεν λέω ότι οι άντρε μερικέ φορές δουλεύουν πλήρη απασχόληση ενώ οι γυναίκες μερική απασχόληση. Όχι, οι γυναίκες μπορεί να δουλεύουν περισσότερες ώρες αλλά οι άντρε δεδομένου ότι δεν έχουν δουλειά στο σπίτι, δεν συμμετέχουν στη, στα παιδιά και στον οικοκυριό, προφανώς έχουν περισσότερο χρόνο για να κάνουν υπερορίε για την έρευνα. Έτσι λοιπόν, οι γυναίκες που είναι μητέρες πάντα αναφέρουν τη δυσκολία συμβατότητας ανάμεσα στη ζωή της μητέρας και της εργαζόμενης, κάτι το οποίο τους δημιουργεί μεγάλο άγχος. Και στην οργανωτική δομή πρέπει να λάβουμε υπόψη μας επίσης το πώς προκυρήσονται οι θέσεις και πώς γίνεται η επιλογή. Πρόκειται για διαγωνισμούς που τελικά δεν είναι τόσο ανοιχτοί στον ανταγωνισμό, ούτε τόσο ανοιχτοί Υπάρχουν διάφορες έρευνες που έχουν γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και η δικιά μου έρευνα δείχνει το ίδιο. Με πολλά παραδείγματα, τα οποία δείχνουν ότι τελικά εκ των προτέρων αποφασίζεται ποιο θα είναι το προφίλ εκείνου που θα πετύχει και αν πρόκειται για προαγωγή πάλι φτιάχνεται η πρόταση για εκδήλωση ενδιαφέροντος με τέτοιο τρόπο, ώστε το προφίλ να είναι συγκεκριμένο. Τώρα, όσον αφορά την ε, ανεπίσημη κατά κάποιο τρόπο οργάνωση, την οτροπία που επικρατεί, την ανεπίσημη δομή της οργάνωσης, αυτή βασίζεται σε σχέσεις, σε πρακτικές, σε συμπεριφορές που οργανώνονται με τέτοιο τρόπο που είναι εχθρικά στοιχεία απέναντι στις γυναίκες. Στην ε, έρευνα στον ακαδημαϊκό κόσμο χρησιμοποιείται και ο όρος μικροπολιτικής. Αυτό ακριβώς σημαίνει ότι παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο οι σχέσεις. Οι σχέσεις μέσα από τις οποίες οι ερευνητές προσπαθούν να προχωρήσουν και να προωθηθούν. Τα παραδείγματα είναι πολλά. Υπάρχουν κοινωνικά δίκτυα που δημιουργούνται μεταξύ εργοδοτών, με άτομα τα οποία έχουν αντίστοιχα χαρακτηριστικά. Όλοι αυτοί φτιάχνουν ένα δίκτυο. Οι γυναίκες δυσκολεύονται πολύ περισσότερο στο να ενταχθούν σε δίκτυα ανδρών. Και επαναλαμβάνω ότι οι άντρε είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν την εξουσία, είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν τι θέσει κύρου συνήθως. Επιπλέον, όταν μιλάμε για μικροπολιτική, μιλάμε και για όλες τις συμπεριφορές εκείνες οι οποίες αποκλείουν γυναίκες. Είτε πρόκειται για ματσισμό, είτε πρόκειται για διακρίσεις. Στοιχεία που είναι παρόντα. Τέλος πρόκειται για τις προσδοκίες και την αξιολόγηση που γίνεται, που βασίζονται στο φύλλο. Δεν περιμένει κανείς η γυναίκα να είναι καλή στη δημόσια ζωή. Αμφισβητείται η ικανότητά της. Οπότε οι απαιτήσει είναι περισσότερες από τις γυναίκες από ότι είναι για τους άντρες. Διεθνείς και ευρωπαϊκές έρευνες και στην Ισπανία, τα δείχνουν όλα αυτά, όπως έλεγα και πριν, χρησιμοποιούνται διαφορετικά κριτήρια ανάλογα με το ποιον θα αξιολογήσουμε. Αλλάζουν τα κριτήρια πρόσληψης ανάλογα με το ποιον θέλουμε να προσλάβουμε. Έτσι λοιπόν η έρευνα δείχνει ότι υπάρχει ανισότητα. Κάθε φορά προσαρμόζονται τα στοιχεία σε αυτούς που θέλουμε να προσλάβουμε ή να προάγουμε. Και γιατί, γιατί είναι οι άντρε αυτοί έτσι καλλιώ που παίρνουν τι αποφάσει και δεν θεωρούν τι γυναίκε ισότιμε με εκείνου. Και γιατί, το λέω αυτό, γιατί του ζητάμε μεγαλύτερη δέσμευση να ανταποκρίνεται περισσότερο σε υποχρεώσει. Αυτό ισχύει και σε θεσμικό επίπεδο και σε επίπεδο νοοτροπίας. Για τις γυναίκες προϋποθέτουμε ότι θα αφιερώσουν περισσότερο τη ζωή τους στη δουλειά τους. Τους ζητάμε περισσότερα προσόντα. Κάτι το οποίο τελικά ε, φροντίζει στο να παραμείνει η διάκριση που γίνεται μεταξύ ανδρών και γυναικών. Τώρα, παρά το γεγονός ότι ορισμένες γυναίκες δεν θέλουν να γίνουν μητέρες και περισσότερες μπορεί να θέλουν να γίνουν μητέρες αλλά δεν θέλουν να παραιτηθούν από τη σταδιοδρομία τους, παρόλα αυτά, αν υπάρχει περίπτωση προαγωγής ή μια νέα θέση, προτιμούν έναν άντρα παρά μια γυναίκα. Και είπαμε ότι επειδή οι άντρε δεν είναι εξίσου υπεύθυνοι για τον οικοκυριό και τα παιδιά, γι' αυτό και είναι περισσότερο στη διάθεση του εργοδότη. Και αυτό είναι πηγή διάκριση. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι γυναίκες είναι μόνο αυτές που γεννάνε, αλλά τόσο οι γυναίκες όσο και οι άντρες γίνονται μητέρες και πατέρες. Το να είναι κανείς πατέρας ή μητέρα όμως δεν σημαίνει το ίδιο πράγμα για μια σταδιοδρομία στη, στα πανεπιστήμια. Προσπάθησα λοιπόν να σας δείξω ότι το φύλλο εξετάζεται σε διαφορετικά επίπεδα. Η κοινωνία πρώτα απ' όλα πρέπει να αλλάξει για να αλλάξει και η κατάσταση στην ακαδημαϊκή σταδιοδρομία. Χρειάζεται αλλαγή και στο θεσμικό επίπεδο και στην οτροπία. Δεν πρέπει να θεωρούμε ότι η γυναίκα είναι το πρόβλημα, ότι η γυναίκα δεν θέλει. Πρέπει να παρέμβουμε στην οργάνωση της ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας που να μην πλήττει τις γυναίκες, που να είναι σε βάρος των γυναικών και να υπάρχει διαφάνεια στις διαδικασίες επιλογής να υπάρχει ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και να μην υπάρχουν πια διακρίσεις ούτε άμεσα ούτε έμεσα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ και θα περάσουμε στα συμπεράσματα στα πλαίσια της συζητήσης μας γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό θεωρώ να συζητήσουμε στο σημείο αυτό να συζητήσουμε πώς ε, θα πρέπει να προχωρήσουμε στη διαδικασία αυτή. Και τώρα θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Πέτεντρελ και μετά το λόγο θα έχει η κυρία Λεγκρίπ για να θέσει ερωτήσεις και φυσικά και οι υπόλοιποι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σε όλους σας. Θα ήθελα να πω ότι σε μεγάλο βαθμό συνάδουν αυτά που είπατε για, με την ανάλυση που έχουμε κάνει και οι τρεις ομιλητές. Είναι συγκλονιστικό να ακούμε τα παραδείγματα που αναφέρετε από τι συνεντεύξει που κάνατε για τι εργασίε. Τα έχουμε ξανακούσει φυσικά βέβαια αυτά. Αλλά είναι νομίζω λογικό το ότι εξακολουθούμε να εντυπωσιαζόμαστε και να θέλουμε να δράσουμε. Θα ήθελα να παραθέσω αυτά που είπατε στην αρχή για το πάθος σας, ότι από την πρώτη στιγμή που ήρθατε σε επαφή με τις επιστήμες ήσασταν ε, ενθουσιασμένοι και από την πρώτη στιγμή εγώ ήμουν ενθουσιασμένος με το ευρωπαϊκό έργο της ενοποίησης και με όλες αυτές τις πτυχές και γι' αυτό λοιπόν η ισότητα των φύλων είναι τόσο σημαντική. Κοιτώντα τη διάσταση της έρευνας και της ανάπτυξης που είναι τόσο σημαντική για την οικονομία μας και για την κοινωνία μας, για την οικονομική και την κοινωνική αξία της. Όσο δεν αξιοποιούμε το πλήρες δυναμικό, το πλούσιο δυναμικό που έχουμε στην Ευρώπη, δεν κάνουμε σωστά τη δουλειά. Και η αλήθεια και η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχουν διαρκείς ανισότητες που επιμένουν και η πρόοδος είναι υπερβολικά αργή. Από τα αριθμητικά στοιχεία που έχω δει στα έγγραφα, τα οποία στέκουν δυστυχώς, δυστυχώς στέκουν. Θα ήθελα να προσθέσω ένα μόνο στοιχείο. 46% είπατε των ε, γυναικών με δεκτορικού, 36% είναι ερευνήτριες 20% είναι κορυφαίες ακαδημαϊκοί και ένα 10% είναι πρίτανης. Το παράδειγμα που ακούσαμε από το Πανεπιστήμιο σας είναι ακριβώς ο μέσος όρος ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν, μία στους δέκα είναι πρίτανης γυναίκα. Είναι και αυτό ένα μεγάλο, μια μεγάλη γυάλινη ροφή. Δεν ξέρω. Τι κάνουμε από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση όμω. Αυτό συνάδει με αυτά που είπατε εσείς κυρία Λόπες ότι προσπαθούμε να φτιάξουμε τις γυναίκες λες και οι γυναίκες ε, είναι το πρόβλημα έχουμε αλλάξει αυτή την προσέγγιση αυτό είναι σημαντικό για να δημιουργήσουμε μια αλλαγή στα θεσμικά όργανα γιατί είναι σημαντικό το πώς τα θεσμικά όργανα αντιμετωπίζουν την ισότητα των ε, φύλων. Άρα έχουμε ένα τρίπτυχο. Καταρχάς θεσμικές αλλαγές. Θα επανέλθω σε αυτό. Κατά δεύτερον, προοπτικές ε, στην καριέρα, στα διαδρομία. Αυτά που είπατε κι εσείς. Και τρίτον, μία πτυχή η οποία ίσως δεν λαμβάνεται επαρκώς υπόψη. Η σημασία της έρευνας βάση φύλου για καλά αποτελέσματα. Πρώτον λοιπόν, θεσμική αλλαγή. Αλλαγή στην ατροπία κατάργηση των εμποδίων. Έχουμε ακούσει κάποια ε, πολιτισμικά ε, εμπόδια. Το παράδειγμα με τον γράφητη που αναφέρθηκε. Ένα εμπόδιο που υπάρχει είναι στη διαδικασία πρόσληψης. Η διαφάνεια λοιπόν στη διαδικασία πρόσληψης είναι πάρα πολύ σημαντική για να υπάρξει ισότητα μεταξύ των φίλων. Τι ζητούμε λοιπόν από τα θεσμικά όργανα και από τα κράτη-μέλη να έχουν σχέδια ισότητας φίλων, Ένας έλεγχος για το πώς έχουν τα πράγματα στα θεσμικά όργανα για την ισότητα των φύλων. Μετά θα συμφωνήσουμε επί των μέτρων και θα τα παρακολουθούμε. Έχει βγουν και βγάζει νόημα. Στην Ευρώπη σήμερα έχουμε μια έρευνα και ξέρουμε ότι περίπου ένα τρίτο των ε, θεσμικών οργάνων έχουν τέτοια σχέδια ισότητας φύλων. Καλό είναι για αρχή, αλλά σε καμία περίπτωση δεν επαρκεί. Δεύτερο στοιχείο για να υπάρχει θεσμική αλλαγή. Χρηματοδότηση. Χρηματοδοτούμε την ανάπτυξη σχεδίων ισότητας φύλου. 70 θεσμούς έχουμε αγγίξει ως τώρα. Είναι σταγόνα στον ωκεανό, αλλά είναι σημαντικό να υπάρξει διάδοση των καλών πρακτικών. Σημαντικό για να πετύχουμε την πρόοδο που θέλουμε. Τέλος. Συνεργαζόμαστε και με τους εμπλεκόμενου φορεί και με τα κράτη-μέλη. Έχουμε ένα project, το οποίο ονομάζεται Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας. Η ιδέα είναι να αξιοποιήσουμε στο βέλτιστο δυνατό βάθμο το δυναμικό που έχουμε στην Ευρώπη και να υπάρξει ελευθερία για τους ερευνητές. Και εδώ είναι σημαντική πτυχή η ισότητα των φύλων πριν από δύο εβδομάδε. ούτε καν, πριν από πιο λίγο χρονικό διάστημα, ομόφωνα τα κράτη-μέλη ενέκριναν έναν οδικό χάρτη για να επιτευθούν οι στόχοι του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και η... τα σχέδια ισότητας φύλων αποτελούν σημαντική πτυχή. Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό στοιχείο για να υπάρξει αλλαγή και να υπάρξει πιο υψηλό ποσοστό από το σημερινό 35% το σημερινό που έχουν τέτοιο σχέδιο ισότητα φύλων. Στον δεύτερο πυλώνα, στη λήψη αποφάσεων. Ξέρουμε ότι οι 18 κράτη-μέλη έχουν ποσοστώσεις για την εκπροσώπηση των υποεκπροσωπούμενου φύλου. Ποσοστώσεις ή στόχους το είπατε και εσείς, ότι υπάρχει νόμος, υπάρχει νομοθεσία, αλλά δεν είναι αρκετά καλή. Το ξέρουμε αυτό και από την νομοθεσία για την ε, ίση αμοιβή, για τους ίσους μισθούς. Ούτε αυτό αρκεί. Χρειάζεται και νομοθεσία και χρηματοοικονομικά κίνητρα και μια πλήρη στρατηγική, ο συνδυασμός όλων αυτών. Και αυτό το ενθαρρύνουμε στα κρατημέλη. Και χρησιμοποιούμε και το βάρος μας ως χρηματοδότες, γιατί υπάρχει ένα όμορφο πρόγραμμα για την έρευνα και την ανάπτυξη με το όνομα Ορίζοντας 2020 και ένα σημαντικό προϋπολογισμό. Και χρησιμοποιείται επίσης για τις ε, προοπτικές σταδιοδρομίας για τις γυναίκες ερευνήτριες. Τα έργα επιλέγονται βάσει αξιολόγησης ομοτύπων. Είναι υψηλός ανταγωνισμός. 10 με 15% μόνο των ε, ετούντων πετυχαίνει. Αν ένα project εκτιμάται στο ίδιο επίπεδο, προτιμάτε το έργο που έχει εκπροσώπηση ισότιμη των φίλων, σε ό,τι αφορά τους ερευνητές που συμμετέχουν. Σημαντικό και αυτό. Επίσης, ζητάμε από τους ομίλους, τους ερευνητικούς που χρηματοδοτούμε να καταθέτουν σχέδια ισότητας φύλων και να το λαμβάνουν υπόψη αυτό το σχέδιο. Γιατί είναι καλό για την απόδοση αυτό. Για την έρευνα φύλου. Αυτή αφορά το να λαμβάνετε υπόψη ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των φύλων στην έρευνα. Αν εργαστούμε, για παράδειγμα, σε θέματα μεταφοράς ε, ηλικιωμένων. Αν δεν λάβουμε και θύλαξης και συγγνώμη, ε, παροχής ε, υπηρεσιών σε ηλικιωμένους, αν δεν λάβουμε υπόψη την διαφορές μεταξύ γυναικών και ανδρών, δεν θα λάβουμε υπόψη ένα σημαντικό παράγοντα του θέματος. Επίσης, πιστεύω ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε, γιατί μιλήσατε και για την εκπαίδευση. Είναι σημαντικό να υπάρχει εκπαίδευση στις θετικές επιστήμες με το να συμμετέχουμε στην πράξη. Με θέματα ισότητας φίλου Και μία τελευταία κουβέντα να πω πριν του περάσω στα συμπεράσματα μου για την επιχειρηματικότητα οι γυναίκες ε, ερευνητέ μπορεί να είναι εντυπωσιακέ ε, επιχειρηματίες. Τα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τις καινοτομίες και τις επιχειρηματικότητα είναι ακόμα χειρότερα από ό,τι στην έρευνα. Και δώσαμε ένα βραβείο σε μια γυναίκα που δημιούργησε μια εταιρεία. Έχει τουλάχιστον 10 υπαλλήλους και κάνει κάτι που έχει να κάνει με την έρευνα. Αυτό το βραβείο λοιπόν δίδεται σε τέτοιες γυναίκες. Έχουμε εκπληκτικά αποτελέσματα. Έχει ξεκινήσει λοιπόν το βραβείο αυτό. Ελπίζω όπως και την προηγούμενη φορά να έχουμε εκπληκτικά αποτελέσματα με γυναίκες ερευνήτριες που παρουσιάζουν τις ιδέες του τα όραματά τους στην αγορά. Άρα, για να ολοκληρώσω, η πρόοδος είναι βαθμιαία. Πρέπει και μπορούμε να κάνουμε πολλά παραπάνω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τις οικονομίες μας. Θα πρέπει να εστιάσουμε σε θέματα θεσμικής αλλαγής και είναι ιδιαίτερα επίκαιρο το θέμα που θίγεται γιατί η επερχόμενη Προεδρία του Συμβουλίου του Λουξεμβούργου έχει θέσει στο πρώτο άτυπο Συμβούλιο που θα διοργανώσει τον Ιούλιο το θέμα της ισότητας των φύλων για να δούμε πώς θα γίνουν αυτές οι θεσμικές οι αλλαγές. Και νομίζω ότι η έκθεσή σας θα αποτελέσει μια σημαντική επιπρόσθετη συμβολή στη συζήτηση και εμείς από πλευρά μας θα χαρούμε να σας δώσουμε επιπρόσθετες πληροφορίες αν το επιθυμείτε. Και για να αναφέρω και τα λόγια του Ζαμονέ, του, του πατέρα ιδρυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μίλησε για θεσμική ε, Ένωση. Τίποτα δεν μπορεί να γίνει χωρίς τους άντρες, αλλά για τους σκοπούς της συνεδρίασής μας θα έπρεπε να έχει πει χωρίς τις γυναίκες, αλλά και τίποτα δεν διαρκεί χωρίς τους θεσμούς. Θα πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε το θέμα της θεσμικής αλλαγής καταπηγόντως. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Σας ευχαριστώ, Λέκη Πρόεδρος. Η κυρία Λεγκρίπ δεν είναι αυτή τη στιγμή στην ε, αίθουσα. Οι Μπορεί μπορούν να πάρουν το λόγο σε περίπτωση που θα ήθελα να πάρει κανείς ε, το λόγο για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Η κυρία Ντανσίλα είναι εδώ στην αίθουσα. Γκούε, η κυρία Βαλίνα, για τους πράσινους, ο κύριος Σεμπαστιάν. Έχετε το λόγο. Σα ευχαριστώ πολύ. Όπω ακούσαμε, σύμφωνα με τις μελέτε και τις πρόσφατε στατιστικές, όλοι συμφωνούμε ότι οι γυναίκε υποπροσωπούνται σε σημαντικούς τομείς ε, της κοινωνικής και επαγγελματικής δραστηριότητας στην έρευνα και την ανάπτυξη, στην επιστήμη, στη λήψη αποφάσεων, σε υψηλόβαθμες θέσεις γενικότερα. Ξέρουμε ότι υπάρχουν χιλιάδες νεαρές γυναίκες οι οποίες έχουν μεγάλο πάθος για την επιστήμη και αντιμετωπίζουν παρόλα αυτά εμπόδια, πολλά εκ των οποίων προ... περιέγραψαν και οι προηγούμενοι ομιλητές. Σύμφωνα με τις πρόσφατες μελέτες, είναι υπερβολικά λίγες οι γυναίκες που ασπάζονται και ακολουθούν μια επαγγελματική ε, επιστημονική σταδιοδρομία. Αυτό οδηγεί σε μια μεγάλη κρίση στην καριέρα τους. Είναι λοιπόν πολύ χαμηλή η εκπροσώπηση των γυναικών και αυτό μας ανησυχεί ιδιότερα σε ό,τι αφορά το επάγγελμα του μηχανικού. Και όπως είπατε υπάρχει αυτό το γυάλινο πλαφόν που εμποδίζει τις γυναίκες, ιδιαίτερα στον τομέα της επιστήμης. Δεδομένου λοιπόν του γεγονότος αυτού και δεδομένου ότι αυτό αποτελεί ένα βασικό ουσιώδες κοινωνικό πρόβλημα και ότι ο άνθρωπος ε, χρειάζεται πιο πολύ παραποτέ την επιστήμη. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, τι στρατηγική πιστεύετε ότι θα πρέπει να εφαρμόσουμε σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση και πώς μπορούμε να προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη προκειμένου να ενθαρρύνουμε τις γυναίκες να ακολουθήσουν μια σταδιοδρομία στον τομέα της επιστήμης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ποιος θέλει να απαντήσει από τους προσκεκλημένους μας. Έτσι. Θα έλεγα ότι είναι μεγάλο το ευρύ το ερώτημα για το πώς μπορούμε να κάνουμε τον προσχετισμό με την εκπαίδευση να αλλάξουμε το μέλλον των γυναικών. Νομίζω ανέφερα ότι ένα από τα βασικά που έχουμε να κάνουμε είναι να βεβαιωθούμε ότι η εκπαίδευση στις θετικές επιστήμες ξεκινά στο δυνατόν νωρίτερα και ότι είναι διαδραστική όπως ανέφερα. Επίσης ότι οι δάσκαλοι και οι καθηγητές κατευθύνονται προ τα διαφορετικά συστήματα καταπολεμώντα το χάσμα μεταξύ των φύλων τη τάξη. Και είναι σημαντικό όταν βλέπουμε ότι έχουμε μια τάξη με αγόρια και κορίτσια, θα πρέπει να μην υπάρχει διαφορετική μεταχείριση. Δηλαδή να μην υπάρχει διάκριση στο φύλλο ε, ε, στην εκπαίδευση. Υπάρχουν διαφορέ στην πραγματικότητα κατά το εκπαιδευτικό σύστημα, στη διάρκεια του εκπαιδευτικού συστήματο που να ενθαρρύνουμε τα κορίτσια να συμμετέχουν περισσότερο λοιπόν οι υπεύθυνοι τη εκπαίδευση πρέπει να το αντιληφθούν και να είναι βέβαιοι ότι όλοι συμμετέχουμε τον ίδιο τρόπο σε μια τάξη. Αυτό είναι ένα στοιχείο που μπορούμε να λάβουμε υπόψη μα ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι ακούγονται όλοι και ενθαρρύνονται με τον ίδιο τρόπο. No, I can only... Απλώς να υπογραμμίσω και εγώ ότι συμφωνώ η εκπαίδευση των ε, δασκάλων είναι σημαντική, εκπαιδεύοντας τους εκπαιδευτές. Έχουμε πολύ ωραίους κύκλους μαθηματών. Ξέρετε ότι οι δεξιότητες δεν είναι απαραίτητα όλες ε, σωστά επεξεργασμένες, αλλά έχουμε πολύ, καλά, πολύ καλούς κύκλους μάθησης, μαθημάτων, για να καταπολεμωθούν οι προκαταλήψεις. Τα κορίτσια χάνουν την αυτοποίθησή του, όπως είπατε. Και ω προ τη φιλοσοφία όμως, σε μια συγκεκριμένη ηλικία αρχίζουν να πιστεύουν ότι δεν είναι καλέ στη φιλοσοφία. Δεν είναι δηλαδή ε, το θέμα των ε, θετικών επιστημών, των STEM όπως λέγονται, ε, επιστήμες, τεχνολογία, οικονομία και μαθηματικά, αλλά και όλα τα υπόλοιπα. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να μοιραστώ και εγώ τις δικές μου προσωπικές μου εμπειρίες και στη Σλοβακία ξεκίνησε, ξεκίνησε αυτό το πρόγραμμα το Λαμάν Αλαπάτε που ανέφερε ο κύριος ε, Ντρουλ και οι φοιτητές, οι μαθητές έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον, πολύ μεγαλύτερο από ότι σε άλλες περιπτώσεις, σε μαθηματικά, χημεία, έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον τα κορίτσια. Είναι μεγάλε οι αποκλήσει όμω μεταξύ των μελών και θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο σε άλλη μια σκιώδη συγγήτρια, στην κυρία Βανίλα Νοβάλ. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Θέλω να ρωτήσω κάτι την κυρία Στρέγια για τα πανεπιστήμια. Γιατί διάβαζα τις προάλλες για μία διάσκεψη της Μαργαρίτα Σάλα, η οποία έλεγε ότι όταν άρχισε την πρώτη ερευνητική της δουλειά, ερευνητική της δουλειά, ο επικεφαλής της, της είπε ότι έπρεπε να της δώσει έναν απλό τομέα επειδή ήταν γυναίκα. Εγώ θέλω να ξέρω γιατί στα πανεπιστήμια θεωρείται δεδομένο ότι οι γυναίκες έχουν λιγότερες ικανότητες ή είναι λιγότερο διαθέσιμες. Μια που δουλεύετε στο Πανεπιστήμιο θα ήθελα να μας πείτε πώς το ζείτε αυτό εκεί. Γιατί υπάρχει αυτή η αντίληψη. Όπως είπα και πριν, μια απάντηση, δεν ισχύει μόνο στο πανεπιστήμιο, γενικά στο κοινωνικό επίπεδο υπάρχουν στερεότυπα, τα οποία συνδέουν τους άντρες και τις γυναίκες με διαφορετικές ικανότητες. Λένε ας πούμε ότι οι γυναίκες έχουμε περισσότερες ικανότητες για ορισμένα καθήκοντα, για ορισμένη σταδιοδρομή, ενώ οι άντρες τα καταφέρνουν καλύτερα αλλού. Έτσι λοιπόν, ενώ στο νοικοκυριό, στο σπίτι και στα παιδιά δεν συμμετέχουν εξίσου άντρες και γυναίκες, αυτό που φτάνει στο πανεπιστήμιο είναι ότι οι άντρες που είναι πανεπιστημιακοί βάζουν τη σταδιοδρομία τους σε πρώτο επίπεδο, ενώ οι γυναίκες βάζουν πρώτα την οικογένειά τους, τα παιδιά τους και μετά την ακαδημαϊκή τους σταδιοδρομία. Ενώ οι άντρες, και ας έχουν και αυτοί παιδιά, είναι παντρεμένοι ή έχουν κάποιους ηλικιωμένους να προσέξουν, να νοιαστούν παρόλα αυτά ότι είναι περισσότερο διαθέσιμοι για τη σταδιοδρομία τους από ότι γυναίκες. Αυτή είναι η δικιά μου εμπειρία. Παρόλο που είμαι νέα ακόμα, το καταλαβαίνω, το διαπιστώνω αυτό κάθε μέρα. Βλέπω τις πιο μεγάλες που κάνουν παιδιά και το βλέπω και στις συνεντεύξεις που έκανα για το διδακτορικό μου. Οι γυναίκες εξηγούν ότι η καριέρα τους προχωράει γρήγορα, η σταδιοδρομία τους προχωράει γρήγορα μέχρι που κάνουν παιδιά. Μετά σταματάει και δεν σταματάει μόνο για την περίοδο που περιμένουν το παιδί τους, αλλά και μετά γιατί δεν τις προσκαλούν τόσο πολύ σε διασκέψεις ή να παρακολουθήσουν κάποια επιμόρφωση. Δεν τις καλούν γιατί θεωρούν δεδομένο ότι δεν θα έχουν αρκετό χρόνο για αυτά. Δεν ρωτάνε τις γυναίκες αν μπορούν να αναλάβουν αυτή την ευθύνη ή όχι. Όχι. Το θεωρούν δεδομένο. Είναι αυτά τα κατεστημένα βάσει των οποίων η γυναίκα είναι λιγότερο διαθέσιμη για πανεπιστημιακή σταδιοδρομία. Σας ευχαριστώ πάρα. Κύριε Σεμπάστια. Ευχαριστώ. Βρήκα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που άκουσα σήμερα το απόγευμα. Παρ' όλα αυτά θέλω να κάνω μια διάκριση. Και αυτά που είπε η δεύτερη ομιλήτρια, που είπε ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε οι άντρε να κάνουν την αλλαγή. Κι όμως, μερικοί από εμά είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε την αλλαγή. Πρέπει λοιπόν να συμμετέχει ολόκληρη η κοινωνία στην προσπάθεια αυτή. Δεν πρέπει να λέμε ότι οι γυναίκες πρέπει να δώσουν τον αγώνα απέναντι στους άντρες. Όντως υπάρχει μια πατριαρχική κοινωνία, αλλά μαζί θα την πολεμήσουμε. Γιατί και οι άντρες ζημιώνονται τελικά. Γι' αυτό το τελευταίο, εγώ πρόσφατα έγινα πατέρας και κανείς δεν θεωρεί δεδομένο ότι χρειάζομαι χρόνο για να είμαι με την κόρη μου. Κανείς. Ξεκολουθώ τον ίδιο ρυθμό στη δουλειά μου και δεν το καταλαβαίνω. Θεωρούν ότι είναι με τη μητέρα της, άρα δεν χρειάζομαι εγώ. Θέλω να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Σίγουρα με ενδιαφέρει πολύ το θέμα, γι' αυτό και ζήτησα από την πολιτική μου ομάδα να είμαι εδώ μέλος. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο τελευταίο ομιλητή, ότι δηλαδή πρέπει να πετύσουμε ποσοστώσει, ότι οι ποσοστώσει είναι ένα μέσο, έτσι δεν είναι αυτό ο σκοπό. Μπορείτε να μα πείτε πιο συγκεκριμένα, παρακαλώ, πώ θα υλοποιηθεί αυτή η πολιτική ποσοστώσεων σε ό,τι έχει να κάνει με το δημόσιο. Για το Πανεπιστήμιο τώρα πιο συγκεκριμένα, στηρίζω το σχόλιο που έγινε για την ε, φιλολογία, φιλοσοφία. Και εγώ είμαι από ένα τέτοιο πανεπιστήμιο και μέχρι την τελευταία χρονιά δεν είχαμε καμία γυναίκα. Το γιορτάσαμε όταν μπήκε στην αίθουσα η πρώτη. Εγώ πήγαινα και παρακολούθησα σύγχρονο χορό και ήμουν μόνο άντρας. Κανένας άντρας άλλος δεν υπήρχε, ήμουνα μόνο εγώ. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιες τέτοιες προδιαγραφές κατά κάποιο τρόπο που εξακολουθούν να ισχύουν. Ζω σε ένα χωριό κοντά στη Βαλένθια, όπου εκεί βρίσκεται το κάμπους των ε, επιστημών. Πράγματι υπάρχει πρόβλημα για θέσεις εξουσίας, αλλά υπάρχει και ένα χειρότερο πρόβλημα. Όταν οι φοιτήτριε παίρνουν το πτυχίο τους και έχουν και καλύτερα ακαδημαϊκά αποτελέσματα, στρέφονται στον ιδιωτικό τομέα, όπου Οι χημικές εταιρείες που έχουμε στην ε, Βαλέθια Αντίθετα, δεν πάνε στον ιδιωτικό τομέα γιατί οι ιδιωτικέ οι εταιρείε, οι επιχειρήσει δεν παίρνουν γυναίκε. Οπότε το μόνο του καταφύγιο είναι το δημόσιο, το πανεπιστήμιο. Θα έπρεπε να τι βοηθήσουμε να μπορούν να περάσουν και στον ιδιωτικό τομέα. Να αλλάξει αυτό. Ξέρω ότι είπα πολλά, αλλά είναι ένα θέμα που βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Δεν πιστεύω ότι οι άντρες έχουν ε, χάσει τη θέση τους ε, στον τομέα των θετικών επιτισμών, των επιστήμων. Δεν μπορώ να πω ότι έχω τέτοια σχετική πείρα. Δεν ξέρω άντρε που να έχουν παραχωρήσει τη θέση του σε μια γυναίκα γιατί θεωρούν ότι κάνει καλύτερα τη δουλειά του. Απλώ θα ήθελα να τονίσω το εξή. Υπάρχουν σχετικέ εμπειρίε στο Πανεπιστήμιο όταν μια γυναίκα λόγου χάρη γίνεται πρόεδρος πανεπιστημίου μετά από τεράστιες προσπάθειες πρέπει να εκλεγεί ο αντιπρόεδρος. Εάν υπάρχουν δύο υποψήφοι, άντρας ή γυναίκα, ε, και η γυναίκα είναι διδάκτορ ενώ ο άντρας έχει απλώς ένα μάστερ, ε, σίγουρα θα επιλεγεί ο άντρας με λιγότερα προσόντα. Δηλαδή, ακόμα και εμεί ω γυναίκε, πρέπει να προσπαθήσουμε να εφαρμόζουμε τα σωστά κριτήρια. Πρέπει να δούμε ποια είναι τα πιο βάσιμα. Και ουσιαστικά είναι το εκπαιδευτικό επίπεδο, είναι κάποιο άλλο στοιχείο. Αυτά είναι γνωστά στην πράξη. Και σε ό,τι φορά το όλο σκέλος της ερώτησης, ίσως να απαντήσει κάποιος άλλος. Και ένα δεύτερο ερώτημα για τις ποσοστώσεις. Yes, for the quotas. Ναι, για τις ποσοστώσεις. Είναι πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα και νομίζω ότι θα μπορούσαν ε, να τεθούν και άλλες ερωτήσεις για τις ποσοστώσεις. Θα ήταν πολύ χρήσιμε και θα μπορούσαμε να δούμε ε, τι πετυχαίνουμε τελικά με τις προσπαθίες μας, οι μεγαλύτερες οργανώσεις, τα ιδρύματα και τα Ινστιτούτα, κάποιες φορές χρειάζονται τέτοιου είδους κινητοποίηση για να μπορέσουν να έχουν ποιότητα και μεγαλύτερη ποικιλία στην πράξη και να μην υπάρχει μόνο η διάσταση του φύλου. Ωστόσο, εγώ ακόμα ονειρεύομαι ότι θα μπορούσε κανείς να πιάσει μια δουλειά και να μην αισθάνεται ότι η ευκαιρία του δόθηκε γιατί ε, υπάρχει ποσόστοση, αλλά ότι ήταν γραφτό του. Αυτό θα ήταν σημαντικό οι εταιρείε λοιπόν να το εφαρμόζουν αυτομάτω και εμεί να το καλύπτουμε ταυτόχρονα στο σύστημα των ποσοστώσεων. Δηλαδή να δίνουμε κατευθυντήριε γραμμέ για το πώ πρέπει όλο αυτό να εφαρμόζεται στην πράξη. Σε κάθε περίπτωση όμω ε, θα πρέπει να επιλέγεται ο σωστό υποψήφιος, το σωστό άτομο για την δουλειά. Δηλαδή, υπάρχει από τη μια ανάγκη να υπάρχει ποικιλία. Ε, σίγουρα έτσι δημιουργούνται καλύτερε ομάδες και μπορούν να γίνουν περισσότερα από αυτά που προσπαθούμε να πετύχουμε στην κοινωνία. Αυτό θα πρέπει να επιδιώκει κάθε οργάνωση οργανισμό. Οι ωστόσο είναι απλώ ένα μέσο. Μέσο να πιέσουμε προ αυτή την κατεύθυνση. Πραγματικά πιστεύω να μην ήταν καν απαραίτητε. Αλλά αυτό παραμένει όνειρο. Πάντως ήταν πολύ καλή ερώτηση. Δεν θα απαντήσω ακριβώς, αλλά θα συνεχίσω με το σχόλιο που έχει να κάνει με τον ιδιωτικό τομέα. Πράγματι, οι γυναίκες τα καταφέρουν καλύτερα στο πανεπιστήμιο, έχουν καλύτερους βαθμούς. Παίρνουν μάστερ, είναι καλύτερα καταρτισμένες. Παρ' όλα αυτά δεν προσλαμβάνονται τόσο πολύ. Σας είπα ποιο είναι τα ποσοστά, ποιες παίρνουν ε, διδακτορικό. Τελικά όμως αυτές που αποφασίζουν για ακαδημαϊκή καριέρα είναι λιγότερες από ότι άντρες. Πριν σας είπα ότι οι διαδικασίες πρόσληψης στο Πανεπιστήμιο μερικές φορές δεν διαπονται από διαφάνεια. Έχω τη δικιά μου επαγγελματική εμπειρία στους ανθρώπινους πόρους και σας λέω ότι στο Πανεπιστήμιο δεν υπάρχει διαφάνεια. Και αν δεν υπάρχει στο πανεπιστήμιο, στον ιδιωτικό τομέα, ακόμα λιγότερο. Όλοι ξέρετε τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στον εργαζόμενο, τον πελάτη. Τελικά οποιαδήποτε επιχείρηση ψάχνει συγκεκριμένα προφίλ εργαζόμενων. Μπορεί να πούνε πιο συγκεκριμένα, μόνο άντρες θέλω. Ή μπορεί να πούνε, διάλεξε τους καλύτερους υποψήφιους και όταν έχουν ε, δύο βιογραφικά αντρών γυναικών, η απάντηση ήταν συνήθως «Μα Αυτά που μα στείλετε μόνο για τους άντρες με ενδιαφέρουν. Οι γυναίκες μένουν σε ενδιαφέρουσα, οπότε δεν με ενδιαφέρουν. Αυτά από την προσωπική μου εμπειρία όταν δούλευα στους ανθρώπινους πόρους. Για το θέμα των ποσοστώσεων. Να σα πω ποια είναι η δικιά μα εμπειρία. Είχαμε θέσει μια ποσόστοση για τη σύνθεση των ομάδων ε, εμπειρογνωμών μας. 50-50-90. Πριν ε, θέσουμε την ποσόστοση αυτή, είχαμε τη φιλοδοξία, αλλά χρειάστηκε η ποσόστοση. Συμφωνώ ότι δεν είναι η καλύτερη δυνατή λύση, αλλά χρειάζεται. Έχουμε και τον ίδιο ποσόστοση για τα πάνελ αξιολόγησης, 60-40% είναι σημαντικό να είμαστε σαφείς, απλοί και να τα συνδυάζουμε αυτά σε εθνικό επίπεδο αυτό που βλέπουμε ότι συμβαίνει, ότι συνδυάζονται στόχοι ποσοστώσεων με κίνητρα, με πολιτικές και κάποια οικονομική υποστήριξη. Από μόνη της η νομοθεσία δεν φτάνει και το βλέπουμε και σε άλλους τομείς και έχουμε και κάποιες ενδιαφέρουσες μελέτες για τη διαφθορά όπου βλέπουμε ότι τα πράγματα δεν φτάχνουν μόνο με την νομοθεσία. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. definovali ako kvóty? Nedalo sa to urobiť proste, že naozaj chcete tam mať vyvážené zastúpenie medzi mužmi a ženami? Že aj pri tak, um, takej malej skupine, ako je napríklad expertná... Και σε μια τόσο μικρή ομάδα όπως μια ομάδα εμπειρογνωμών χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε ποσοστώσεις. Έχασα τη μετάφραση, λέει ο μου Η ερώτησή μου είναι αν έχετε πραγματικά ανάγκη από ποσοστώσεις στην ομάδα εμπειρογνωμών ή αν θα μπορούσε να υπάρχει μια μικρή ομάδα Είναι σαφές η εμπειρία μας, μας δείχνει το εξή ότι δεν ξέρω κατά πόσο αυτό έχει να κάνει με τα λόμπι, γιατί αναφερθήκατε στα λόμπι. Ναι, υπάρχουν λόμπι. Το θέμα είναι η εξουσία και η επιρροή. Υπάρχει το λόμπι των ανδρών, ναι. Λέει πρόεδρος. Η δική μας εμπειρία είναι το εξή ότι πάντα υπάρχουν επιχειρήματα. Ότι υπάρχει ένας άνδρας, ότι το προφίλ δεν ξέρουμε αν είναι καλό. Υπάρχει μια έλλειψη ροής ε, στο σύστημα αυτό. Και αν θέλουμε να είμαστε στο σύστημα αυτό πρέπει να είμαστε πολύ σαφείς ε, και ξεκάθαροι, η Πρόεδρος. Τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Σόιντροβα και μετά στην κυρία Λεγκρίπ. Ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις σας, για τη συμβολή σας. Ήθελα να προσθέσω κι εγώ μερικές σκέψεις. Πιστεύω ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των χωρών και υπάρχουν και διαφορετικές εξελίξεις. Η κυρία Λόπες μας είπε ότι στην Ισπανία και την Πορτογαλία 40% των γυναικών ενδιαφέρονται να πάρουν πτυχίο πανεπιστημίου ε, και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Στην Δημοκρατία της Τσεχίας 60% των γυναικών ε, φοιτούν στα πανεπιστήμια ως φοιτήτριες. Ε, οι γυναίκες δηλαδή έχουν τα προσόντα, είναι έξυπνες, έχουν τη διάθεση και θέλουν να, έχουν, να πάρουν πτυχίο. Όμως μετά Μετά τα 27 αλλάζουν τα πράγματα. Δηλαδή γίνονται μητέρες. Η μητρότητα είναι σε ένα βαθμό και θέμα μίμησης αλλά και θέμα προνομίων. Πρέπει λοιπόν να βρούμε τον τρόπο να στηρίξουμε τις γυναίκες για να μπορούν να συνεχίσουν την καριέρα τους ως ακαδημαϊκοί στο Πανεπιστήμιο και ως επαγγελματίες στα πανεπιστημιακά ιδρύματα και στις θετικές επιστήμες. Ευχαριστώ τον κύριο Ντρόλ γιατί πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματικά επιδιώκει να βρει πρακτικά μέσα για να στηρίξει την συμμετοχή των γυναικών στα ερευνητικά ιδρύματα, σε ομάδες εμπειρογνωμόνων. Τα παραδείγματα που δώσατε τα κατανοώ πάρα πολύ καλά και κατανοώ γιατί επιλέξατε αυτές τις ποσοστώσεις για αυτά τα προγράμματα, για αυτούς τους διαγωνισμούς, γιατί είναι προφανές, είναι ξεκάθαρο Νομίζω ότι είναι πιο πρακτικό. Ε, και μάλλον και αναγκαίο σε αυτό το τομέα. Επίση, αυτό που είναι επίση σημαντικό είναι ότι στην Δημοκρατία τη Τσεχία τα πανεπιστήμια άρχισαν να προβλέπουν παιδικού σταθμού, νηπιαγωγεία, για να μπορούν οι καθηγήτριες, οι γυναίκες καθηγήτριες, αλλά και οι φοιτήτριες να ξέρουν ότι μπορούν να φροντίσουν τα παιδιά τους. Πρέπει να βρούμε και τα απαραίτητα οικονομικά μέσα βέβαια να στηρίξουμε τις γυναίκες στους ε, ρόλους αυτούς, στην ακαδημαϊκή τους καριέρα. Και στο τέλος, εν τέλει θέλω να πω και το εξής. Οι ποσοστώσεις για τα πανεπιστήμια δεν είναι κάτι που μπορεί να εφαρμοστεί λόγω της ακαδημαϊκής ελευθερίας. Είναι αδύνατο. Τα πανεπιστήμια ψηφίζουν τους πριτάνεις, τους καθηγητές και ούτω καθεξής. Βεβαίως αυτό που μπορούμε να αλλάξουμε και που μπορούμε να ασκήσουμε επιρροή είναι η στάση των κυβερνήσεων και των ε, ηθινόντων, δηλαδή τα διοικητικά συμβούλια και τα ελεγκτικά συνέδρια στις διάφορες χώρες ανάλογα με την νομοθεσία του. Στον τομέα αυτό έχουμε τη δυνατότητα Euh, Μπορούμε να βοηθήσουμε τη συμμετοχή ε, των γυναικών ακαδημαϊκών που να είναι stakeholders για την διαχείριση των πανεπιστημίων ε, και των θετικών επιστημών στα κάτι μελη Ευχαριστώ πολύ για την προσέγγισή σας. Να προσθέσω και εγώ ένα στοιχείο. Αυτό που προβάλλατε είναι η ανάγκη να υποστηρίξουμε τις γυναίκες στην φάση που κάνουν παιδιά προκειμένου να μπορέσουν να συνεχίσουν γιατί σε πολλά πανεπιστήμια είναι πολλές οι γυναίκες ε, που συμμετέχουν αλλά η συνέχεια στη σταδιοδρομία τους είναι το θέμα. Γι' αυτό λοιπόν ε, μία από τις προτάσεις που έκανα αντί να κοιτάμε τις άδειες μητρότητες, να το κοιτάξουμε ως άδεια οικογένειας, ε, κάτι που να δικαιούται και ο άντρας και η γυναίκα. Νομίζω ότι από πλευράς οικογένειας θα πρέπει να το κοιτάξουμε έτσι. Υπάρχει μεγαλύτερη ισότητα, πιο ίσια, ίση συζήτηση μεταξύ ανδρών και γυναικών όταν υπάρχει μια καινούργια οικογένεια. Είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι μεταξύ γυναικών και ανδρών υπάρχει μια ίση κατάσταση. Αυτό που συμβαίνει συχνά είναι ότι οι γυναίκες αποτρέπονται από το να ακολουθήσουν μια σταδρομία όταν κάνουν παιδιά. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Ρεγκρίπ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, Ζητώ συγγνώμη εκ μέρου τη καθήλυνη συγκεντρία τη κυρία Βόζεμπερκ, που δεν μπορεί να είναι παρούσα. Έκθεση ιδία πρωτοβουλία τη Επιτροπή Γυναικών, συναρπαστικότατη. Και καινοτόμα. Και εγώ να ζητήσω συγγνώμη γιατί δεν μπόρεσα να είμαι ούτε εγώ εδώ έπρεπε να ψηφίσω σε μια άλλη επιτροπή. Δυστυχώς αυτή είναι η μοίρα μας εδώ στο Κοινοβούλιο. Θα ε, έπρεπε να, να διεξαγάγω κάποια συμπεράσματα για, για παρεμβάσεις τις οποίες δυστυχώς δεν άκουσα καθόλου ολοκληρία, οπότε αυτό είναι κάπως ακροβατισμός, αλλά οι προτάσεις σας και οι τοποθετήσεις σας νομίζω είναι, ήταν κέρυες, το είπαν οι συνάδελφοι ε, στις παρεμβάσεις σας με τις διαπιστώσεις, με τις διαγνώσεις, με τις προτάσεις, με τις συστάσεις σας που ήταν ακριβέστατες και πολύ συγκεκριμένες. Πέραν όλων αυτών πρέπει να πάρουμε κουράγιο και να πούμε τρεις κουβέντες για να δούμε πώς μπορεί να διαρθρωθεί η έκθεση η οποία θα ψηφιστεί. Σε αυτή τη φάση η κυρία και η συγγητριά μας και οι σκιώδες εισηγητές της Επιτροπής έχουν ήδη ετοιμάσει ένα πρώτο ε, σχέδιο γράφου για να συζητήσουν μεταξύ τους. Νομίζω ότι ήταν μια καλή βάση εργασίας. Ε, θα είναι πραγματικά ε, πλούσια η ανταλλαγή απόψεων. Τι ερχόμενε εβδομάδε θα συζητήσουμε το θέμα τη αυτοπεποίθησης, τη εργασία και του εθελοντισμού. Θα πρέπει να τα δούμε αυτά σε έναν ορίζοντα μακροπρόθεσμο αλλά και βραχυπρόθεσμο. Δηλαδή τι μπορούμε να κάνουμε τώρα εδώ, τι μέσα διαθέτουμε για να, ε, για να ακολουθήσουμε αυτές τις τρεις, αυτούς τους τρεις φάρους, αυτές τις τρεις σημαδούρες, αυτούς τους όρους που σαν στίγμα θα πρέπει να καθοδηγήσουν ε, την πορεία μας στον ορίζοντα. Τα νεαρά κορίτσια δηλαδή, μεγαλώνοντας, γίνονται πιο έξυπνα, πιο σοφά, αλλά με τα στερεότυπα, τους φραγμούς που έχουν να αντιμετωπίσουν, τις αόρατους φραγμούς που ε, τελικά βαρύνουν, βαρύνουν τους ώμους μας και υπονομεύουν υποσκάπτουν την αυτοπεποίθησή μας σε αυτή την περίπτωση. Βλέπουμε ότι η ελίτ, η ε, ταγή της κοινή γνώμης, οι εκπρόσωποι των, ε, ε, του πνευματικού κόσμου χρειάζονται την ενέργεια των γυναικών αυτή, που είναι θαυμάσια, τα κορίτσια και οι γυναίκες στην Ευρώπη, με τόσο υψηλά προσόντα, με τόσο πολύ μεγάλη συμμετοχή στα πανεπιστήμια και τις επαγγελματικέ σχολές, δεν έχουν τόσο υψηλή, τόσο έντονη παρουσία, και αυτό είναι ένα από τα βασικότερα σημεία της έκθεσης, στις τεχνικές και επαγγελματικές και επιστημονικέ σχολέ. Πρέπει να ανακτήσουν οι γυναίκε την αυτοπεποίθησή του. Πρέπει να ανακτήσουν την, την πίστη του στο σύστημα. Οι εκπαιδευτέ, το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να ε, δώσουν διαφορετικό ρόλο στις γυναίκε, να μπορούν να εξοικειωθούν με την γνωσία των επιστημών, τη τεχνολογία, να ξεπεράσουν τα στερεότυπα, τα κλισέ, ένα σωρό πράγματα που κάποιες φορές ε, κάποιες φορές είναι ε, δυστυχώς αόρατα εμπόδια για τις ανθρώπινες σχέσεις και μας ε, προκαταβάλουν ως προς τη συμπεριφορά μας και ως, και ως προς την εκπαίδευση. Εμείς ως μπαμπάς και ως μαμά θα πρέπει να προσέξουμε τι κάνουμε για τα κορίτσια μας ώστε το εκπαιδευτικό σύστημα, η κοινωνία στο σύνολό της τα οπτικοακουστικά, τα σχολικά βιβλία, οι ε, πολιτιστικές ε, ενώσεις. Ότι ε, είναι ουσιαστικά ε, παρόν στην καθημερινότητα των κοριτσιών μας μπορεί να επηρεάζουν ε, τα μυαλά των νεαρών παιδιών. Θα πρέπει λοιπόν το στοιχείο της εκπαίδευσης να είναι ένα εργαλείο που θα χρησιμοποιηθεί ώστε να μπορούμε να ξεπεράσουμε τις προκαταλήψεις, τα στερεότυπα και να τα καταπολεμήσουμε με κάθε τρόπο. Χρειάζεται λοιπόν και η εθελοντική δράση από την πλευρά των πολιτικών ευθυνόντων, των οικονομικών φορέων. Ε, εμείς, εμείς το Κοινοβούλιο με την έκθεση αυτή ελπίζω ότι θα είμαστε σε θέση να επηρεάσουμε τα πράγματα. Μπορούμε να κάνουμε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις με συγκεκριμένα μέτρα από την θετική διακριτική διακριτική μεταχείριση μέχρι τις νομοθετικές προτάσεις. Θα δούμε. Θα δούμε. Θα είναι αντικείμενο τη συζήτησης μεταξύ των ομάδων. Αλλά χρειάζονται πολύ συγκεκριμένα χειροπιαστά μέτρα και να υπάρχει πραγματικά διάθεση από την πλευρά όλων. Η ισότητα λοιπόν είναι ένα θέμα. Εδώ είμαστε στην ε, Επιτροπή των Δικαιωμάτων των Γυναικών. Υπάρχει θέμα δικαιοσύνη, ισορροπίας, αρμονίας Ε, των κοινωνιών μας που πρέπει να προσπαθήσουμε να τις βελτιώσουμε για να φτάσουν στις σωστές συνειδητοποίησεις. Και βεβαίως υπάρχει και αυτή η μεγάλη σπατάλη. Βλέπουμε τους γυναικείους πόρους, για να τους ονομάσω έτσι, την ενέργεια των γυναικών να μην αξιοποιείται πλήρως. Στην επαγγελματική πορεία που μπορεί να δίνει ε, αξία στις γυναίκες για να ανέβουν τα κλιμάκια της ιεραρχίας και νομίζω ότι για το μέλλον των κοινωνιών μας είναι σημαντικό η έρευνα, οι επιστήμες, η ακαδημαϊκή εργασία, όλα αυτά να σφυριλατήσουν το χαρακτήρα της μελλοντικής κοινωνίας. Εκεί που θα ζήσουμε, που θα ζήσουν τα παιδιά μας, τα παιδιά των παιδιών μας. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε την ενέργεια και το δυναμικό των γυναικών. Πρέπει να ε, κάνουμε ό,τι μπορούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει να ανακτήσουμε την αυτοπεποίθησή μας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε σε αυτή την ομάδα, αλλά πραγματικά οι Σκιώδης και η κυρία Βόζεμπεργκ θα ε, συμβάλλουν προς αυτόν τον κοινό σκοπό με όσα ακούσαμε σήμερα το απόγευμα και βεβαίως σας έχουμε εμπιστοσύνη για να διορθώσετε τις ε, κατάλληλες προτάσεις για την αυτοπεποίθηση, την παιδεία και ε, την ε, σωστή επιλογή των προτάσεων. δυστυχώς δεν άκουσα όλες τις παρουσιάσει, αλλά πρέπει να πω το τελευταίο πράγμα που ήταν πολύ χαρακτηριστικό ήταν η κρυστάλλινη ροφή και ο λαβύρινθο που ε, αναφέρατε. Μία περιγραφή πραγματικά ε, πολύ γλαφυρή ε, με όλη την αγωνία που μπορεί να ε, κρύβει ένας λαβύρινθος. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα μπορούσαμε να το αναπτύξουμε πολύ περισσότερο το θέμα αυτό να υπενθυμίσω ότι στις 15 και 16 Ιουνίου θα συζητήσουμε την έκθεση αυτή. Ε, τότε λοιπόν ε, μπορούμε να συζητήσουμε και σε επίπεδο σκιωδών. Δεν ξέρω αν θέλετε να πάρετε πάλι το λόγο, αγαπητοί ομιλητές, να κλείσουμε. Ναι. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσουμε για το θέμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι αν συνεργαστούμε πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε διαφορά. Όπως ανέφερα και στο τέλος, μου άρεσε και εμένα η ιδέα της κρυστάλλινης οροφής. Γιατί το γυαλί μπορούμε να το σπάσουμε εύκολα. Πολλά λοιπόν μπορούμε να κάνουμε αν συνεργαστούμε και μάλιστα με τρόπο για να σημειώσουμε μεγάλη διαφορά. Αυτό το θέμα το έχω συζητήσει πραγματικά τόσο πολύ καιρό για υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα. Σας ευχαριστώ. Να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω όλους τους αρμόδιους που μας άκουσαν και προφανώς πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να σπάσουμε αυτό το αόρατο πλαφόν, αυτό το, την αόρατη οροφή και να σημειώσουμε τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των ανθρώπων. Αυτός ήταν ένας τρόπος να καταρρύψουμε αυτά τα εμπόδια που υπάρχουν. Θέλω να ευχαριστήσω για τα σχόλια που ακούσαμε και όλοι σας να συνεχίσετε να δουλεύετε πάνω σε αυτό το θέμα. Εννοείται ότι η κατάσταση της γυναίκας βελτιώνεται σιγά σιγά και στις επιχειρήσεις και στα πανεπιστήμια και στην κοινωνία. Μένουν όμως πολλά ακόμα να γίνουν. Γι' αυτό θέλω να σας ενθαρρύνω να συνεχίσετε. Πιστεύω ότι έχουμε στην Ευρώπη την παράδοση και το δυναμικό να κάνουμε τη διαφορά γιατί μπορούμε να αναπτύξουμε πολλές καλές πρακτικές, να αναπτύξουμε πολλά μοντέλα, εκπληκτικά μοντέλα. Μαζί λοιπόν αναμένει μπορούμε να τα πετύχουμε αυτά. Σας ευχαριστώ λέει Πρόεδρος. Θα ευχαριστήσω τους αξιότιμους προσκεκλημένους και θα δώσω το λόγο τώρα στην κυρία Σαμπόσκα για το σημείο 21, για την έκθεση, για την εφαρμογή της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για την ενοποίηση της αρχής ε, της ισότητας ε, γυναικών ε, και ανδρών στα θέματα απασχόλησης. Ευχαριστώ πάρα πολύ, συνάδελφοι. Θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω όλους και όλες για την συνεισφορά σας για την έκθεση αυτή. Έτσι όπως έχουν τώρα τα πράγματα, έχουμε 169 τροπολογίες με στόχο να βελτιωθεί το σχέδιο κειμένου, το σχέδιο έκθεσης δηλαδή, όσον αφορά την εφαρμογή και την ε, διατύπωση της εφαρμογής της οδηγίας του 2006 σχετικά με την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης. Έχοντας διαβάσει όλες τις τροπολογίες, είμαι ειλικρινά ευγνώμων απέναντί σας για την ενεργό συμμετοχή σας. Επιτρέψτε μου όμως να κάνω κάποια σχόλια σχετικά με τις τροπολογίες αυτές. Οι περισσότερες από τις τροπολογίες που διάβασα θα έλεγα ότι ανήκουν σε τρεις κυρίως κατηγορίες. Ποιες είναι αυτές, πρώτον. Αυτές που έχουν ως στόχο να διευκρινίσουν ακόμα περισσότερο το κείμενο. Και γραμματικά και συντακτικά, αλλά και να το καταστήσουν νομικά πιο σαφές. Η δεύτερη κατηγορία είναι τροπολογίες που προτείνουν νέα μέτρα για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών. Εδώ θα ήθελα να μνημονεύσω ιδιαίτερα τις προτάσεις που αναφέρονται σε κυρώσεις σε βάρος των εργοδοτών εκείνων οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με την αρχή αυτή της ίσης μεταχείρισης όταν πρόκειται για ίδιας αξίας εργασία. Και πρόκειται και για ευκολία πρόσβαση στη δικαιοσύνη μέσω μιας δικαστικής αρρωγής ή μέσω μεγαλύτερης συμμετοχής των συνδικάτων, των μη κυβερνητικών οργανώσεων και των τοπικών αρχών. Μ' αρέσει επίσης πάρα πολύ η πρόταση που λέει να υπάρξει ένα ευρωπαϊκό έτος καταπολέμησης των διαφορών στους μισθούς μεταξύ ανδρών και γυναικών στο βαθμό που ειλικρινά πιστεύω ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ακόμα περισσότερο, το ευρυκοινό δηλαδή, ότι υπάρχει αυτή η διαφορά. Η τρίτη και τελευταία κατηγορία αποτελείται από τροπολογίες που θα τις ονόμαζα ιδιαίτερα φιλόδοξες, επειδή προσπαθούν να εντοπίσουν τι αιτίε της ανισότητας και να δούμε ποιοι είναι οι κοινωνικοί παράγοντες εκείνοι που συνεισφέρουν στην ανισότητα αυτή. Οι τροπολογίες της τρίτης αυτής κατηγορίας αναφέρονται για παράδειγμα στην βία σε βάρος των γυναικών, στη μητρική, μάλλον στην άδεια μητρότητας, πατρότητας, στις διακρίσεις που γίνονται σε βάρος των ατόμων με αναπηρίες ή ειδικών αναγκών. Δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι μπορούμε να έχουμε πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για όλα αυτά τα θέματα, αλλά πρέπει να σας πω ότι ε, φοβούμε για τις τροπολογίες αυτές αν συμπεριληφθούν στην ε, έκθεση. Γι' αυτό θα ήθελα να πείσω κάποιους από εσά, των οποίων οι τροπολογίες ανήκουν στην κατηγορία αυτή, να ξανασκεφτούν τις τροπολογίες τους και ενδεχομένω να τις αποσύρουν εάν πιστεύετε ότι όντω ξεπερνούν τα πλαίσια της οδηγίας αυτής. Αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρομαι εκ των προτέρων, μπορώ να σας πω, που μπορώ να συνεργαστώ μαζί σας για συμβιβαστικές τροπολογίες. Είμαι ανοιχτή στις προτάσεις σας, γιατί ειλικρινά πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε στο τέλος ένα κείμενο που θα υποστηρίξουν οι ευρωβουλευτές από όλες τις πολιτικές ομάδες. Μαζί μπορούμε να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα. Όταν πρόκειται για απασχόληση, η ανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι κάτι που δεν μπορούμε να ανεχτούμε. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα θα δώσω το λόγο στους άλλους ευρωβουλευτές. Με πρώτη την κυρία Ντέλη. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ω ε, σύνηση σκιώδη εισηγήτρια, θέλω να πω στην κυρία Ζαμπόρσκα ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την αφοσίωσή σας, για την επιμέλεια που προβλέψατε αυτήν την περιβόητη οδηγία του 2006 στην ε, συζήτησή μας και που κάνατε αυτή τη δουλειά, δουλειά που είναι σχολαστική, γιατί επιμένετε στις λεπτομέρειες, σε όλες τις πτυχές της οδηγίας. Όντως θα πρέπει να ε, γίνει εδώ ένα brand fair, διότι η Επιτροπή των Γυναικών δεν πρέπει να παραμείνει απλώς γυναικεία επιτροπή που δημιουργεί μια σωρία εκθέσεων. Όχι. Η έκθεση αυτή δεν πρέπει να, γίνει, να είναι μια έκθεση που θα παραμείνει στα χαρτοκούτια και θα βγαίνει κάθε δύο χρόνια όταν θέλουμε να τη θυμηθούμε. Θα πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι η έκθεση αυτή ζητά με σαφήνεια την μεταφορά που ω τώρα ήταν πλημελή από τα κράτη-μέλη τη οδηγία αυτή. Αυτό είναι ο στόχο μα. Να πούμε ότι δεν μπορούμε πλέον να μείνουμε στην κατάσταση ω έχει, γιατί ε, κατεπήγει ε, η επίλυση του προβλήματο. Νομίζω ε, ότι έχουμε φτάσει πια στο 2015 και μιλάμε ακόμη για μισθολογική ανισότητα που δεν δικαιολογείται. Εδώ βλέπω την ε, ε, προσπάθεια που έχουν κάνει ως τώρα η γιαγιά μου, η μάνα μου και η δική μου γενιά έχει να αντιμετωπίσει τα ίδια προβλήματα. Πρόκειται για ένα βασικό πρόβλημα των γυναικών μετά από 40 χρόνια νομοθεσίας. Και βλέπουμε ότι πρόοδος έχει γίνει. Πρόοδος όμως που για την ώρα είναι αρκετά ε, ανεπαρκής. Οι αριθμοί το λένε. Είναι τεράστιο το χάσμα πληρωμών. Ε, θα ήταν ωραίο λοιπόν στην ε, έκθεσή σας, επειδή τονίζετε το γεγονός ότι οι γυναίκες είναι θύματα αυτής της κάθετης διάκρισης αλλά και οριζόντιας διάκρισης, να ε, θυμόμαστε ότι δεν χάνουν μόνο το μισθό τους, αλλά επειδή ξέρω ότι έχετε μεγάλο ενδιαφέρον για όλο αυτόν τον αγώνα, αυτή την προσπάθεια, μην ξεχνάμε τον υπολογισμό των συντάξεων, κάτι που δεν είναι αμεληταίο. Ε, παρά το γεγονός λοιπόν, και εδώ θα σας στηρίξω, Πρέπει να ε, ζητήσουμε μελέτες, πρέπει να ζητήσουμε να γίνουν έρευνες, να ζητηθούν καλές πρακτικές, ε, να αναλάβουμε τις σωστές πρωτοβουλίες, ε, πηγαίνοντας προς τη σωστή κατεύθυνση γιατί χωρίς δεδομένα, χωρίς πληροφορίες δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τους αρχικούς κρατών και κυβερνήσεων. Αυτοί έχουν το κλειδί της επιτυχίας στα χέρια του. Και Βλέπουμε τι είδου διακριτική μεταχείριση μπορεί να επιβληθεί στις γυναίκες. Εδώ ε, πρέπει να θυμίσω μια σειρά από τροπολογίες ότι πρέπει να παρέμβουμε και με την εκπαίδευση. Ε, πρέπει να πάυσουν τα στερεότυπα να ισχύουν, να μην ε, υπάρχουν τέτοιες προκαταλήψεις κατά των γυναικών σε επιστημονικούς κλάδους και εκπαιδευτικούς κλάδους που επιφυλάσσονται μόνο στους άντρες που ε, διαπρέπουν μόνο οι άντρε, να θυμίσω αυτό που λέγαμε πριν για τις θετικές επιστήμες εδώ υπάρχει μια πραγματική πρόκληση για τις γυναίκες Διότι νομίζουμε ότι η εκπαίδευση στις θετικές επιστήμες ξεκινά μόνο στο σχολείο. Όχι, όχι. Ε, αυτό αρχίζει και γίνεται και στην εξουσχολική ε, κατάρτιση και εκπαίδευση. Γι' αυτό έχω υποβάλει τροπολογίε που αναφέρονται σε αυτές τις διακριτική, μορφές διακριτικής μεταχείρισης κατά πολλών ε, προσώπων λόγω του φύλου. Οι λόγοι της διακριτικής μεταχείρισης είναι πολλοί και καλό είναι να δούμε και την μερική εργασία, ένα πρόβλημα ξεκάθαρα γυναικείο, το αποδεικνύουν οι αριθμοί. Οι γυναίκες σήμερα δεν είναι απλώς γυναίκες, πρέπει να ε, αναλάβουν όλες τις δυσκολίες ενός επαγγελματικού πεδίου, να αναλάβουν νέα καθήκοντα και ως προς αυτό ε, έχουν τεράστιες ευθύνες. Όλα αυτά είναι αρκετά δυσβάσταχτα. Δεν έχουν συμπεριληφθεί στους υπολογισμούς μας. το απολογισμό του ΑΕΠ δεν ε, καταδεικνύεται από τους δείκτες της, ε, του πλούτου. Οι γυναίκες κάνουν πάρα πολλά. και βλέπω μας μιλάνε για τους, ε, ε τους γονιούς τους, για τους προγονούς τους οι γυναίκες. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για την κοινωνία, γιατί χωρίς αυτά τα εισοδήματα δεν μπορεί να υπάρξει κοινωνική πρόοδος. Οπότε στο μεγαλύτερο μέρος των μονογονεϊκών οικογενειών, όπου ο μόνος γονέας είναι γυναίκα, ε, υπάρχουν και δραματικές συνέπειες για τις συνθήκες διαβίωσης των γυναικών. Οι συνθήκες αυτές η σύνθεση μιας οικογένειας είναι μια πολύ σημαντική πτυχή. Έπειτα, το ξαναλέω, αλλά πραγματικά πρέπει να δοθεί τέρμα στη μισθολογική διάκριση. Θα πρέπει πραγματικά σήμερα οι διακρίσεις ε, να σταματήσουν. Μπορεί οι δύο θέσεις να ε, είναι ακριβώς οι ίδιες στην περιγραφή τους, αλλά να αλλάζει το κύριο και κυρία μπροστά από το όνομα. Ε, Πρέπει να σταματήσει αυτή η διακριτική μεταχείριση, δηλαδή ίση εργασία, ίσω μισθός. Και είναι πάρα πολύ εύκολο να αλλάζει ε, ε, ο χαρακτηρισμός μιας θέση για να πληρώνεται λιγότερο μια γυναίκα. Υπάρχουν επιχειρήσεις που πραγματικά αλλάζουν τον τίτλο ενώ πρόκειται για τα ίδια καθήκοντα, ώστε η γυναίκα να πληρώνεται λιγότερο. Και αυτό λοιπόν πρέπει να το τονίσουμε. Επίσης σήμερα Πρέπει να έχουμε και κάποια κριτήρια για να συγκρίνουμε μεταξύ τους τις θέσεις εργασία. Το ζητάει και η έκθεση η έκθεση θα πρέπει να εκπονήσει έναν οδηγό με ένα σύστημα αξιολόγησης, ουδέτερης αξιολόγησης των επαγγελματικών κλάδων και νομίζω ότι όλα τα κρατημέλη πρέπει οπωσδήποτε να προβλέψουν ένα τέτοιο σύστημα. Διότι πραγματικά θα μπορούσαμε έτσι να εντοπίσουμε ποιε είναι οι, οι μορφές διακριτικής μεταχείρισης, είτε έμεσες είτε άμεσες. Και νομίζω ότι υπάρχουν και συγκεκριμένα στοιχεία που μπορούμε να προσκομίσουμε στη δικαιοσύνη για να εντοπίσουμε τις μισθολογικέ αποκλήσεις και αυτό θα μας, ε, μπορούσε να μας αποφέρει σημαντικά πραγματικά ωφέλη. Επίση, να δούμε και το θέμα τη διαφάνεια ε, στο σύστημα της, ε, το μισθολογικό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη έχει προτείνει μέτρα από το 2014 με τι συστάσει τη, με την ε, νέα νομοθετική πρόταση, με την κατάρτιση των μισθωτών, με τι ελέγχου των μισθών. Και σωστά το θυμήσατε, κυρία Ζαμπόρσκα, θα πρέπει πραγματικά να κάνει τα πάντα και να προτείνει ό,τι καλύτερο μπορεί για τα πρόστιμα. Πρέπει να πιέσουμε τις επιχειρήσεις να σεβαστούν τον κανόνα της ε, ισότητας, ε, της μισθολογικής ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ε, εγώ δουλεύω και στην Επιτροπή Μεταφορών. Οι αεροπορικές εταιρείες όταν δεν ακολουθούν τα σωστά κριτήρια μπαίνουν σε ένα μαύρο κατάλογο και κάνουν τετραπλές προσπάθειες μετά για να βγουν από αυτόν τον μαύρο κατάλογο. Ε, ε, θα έπρεπε λοιπόν μάλλον να έχουμε ένα μαύρο κατάλογο ε, για να κάνουν οι εταιρείε αυτό που πρέπει. Και θα πρέπει να το πούμε με τρόπο απλό και εύληπτο. Μ' αρέσει η κυρία Ζαμπόλσκο ο ρόλο που προβλέπεται για του κοινωνικού εταίρου, για τι μη κυβερνητικέ οργανώσει και θα πήγαινα ακόμη μακρύτερα Νομίζω ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη ε, σημασία και στους εθνικούς οργανισμούς πρόθεση της ισότητας, της ίσης μεταχείρισης. Είναι πολλοί οι οργανισμοί στα διαφορα κατημέλη, είναι ανεξάρτητοι και ε, πρέπει να δούμε τις μισθολογικές πρακτικές, ε, το κατά πόσον οι γυναίκες μπορεί να έχουν εύκολη πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Όλα θα τα βρίσκουμε στην έκθεση και τέλος και θα ολοκληρώσω, Πρόεδρε, διότι είπατε ότι μιλάω πολύ, αλλά είναι ένα θέμα που μας παθιάζει. Αυτό που ζητούμε εμείς είναι τα κράτη-μέλη να αναλάβουν τις ευθύνες τους ως οικολόγια και πράσινοι. Θα πρέπει να είμαστε εδώ υποδηματικοί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν πολύ σαφής. Δεν μπορεί να μας παραπέμψει σε αυτά που θα γίνουν σε μια διετία, τριετία και το Ε, πρέπει η Επιτροπή να προβλέψει δεσμευτικά μέτρα με στόχους, με ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, διότι καθόλου δεν θέλω να τελειώσει η θητεία μου όπως έγινε την πρώτη φορά και πάλι να πούμε ότι δεν καταφέραμε τίποτα. Θα πρέπει να έχουμε μια θητεία και το είπε ο κ. Γιούνκερ, ήταν η τελευταία ευκαιρία της, ευκαιρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα λοιπόν να δούμε ε, εάν δεν έχουμε και την τελευταία ευκαιρία για την ισότητα ανδρών και γυναικών. Euh, Ευχαριστούμε. Η κυρία Μπέρντερ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ Σας πολύ. ευχαριστώ πολύ. Πολλά από αυτά που από αυτά που ήθελα να πω ήδη έχουν καλυφθεί. Θα ήθελα όμως στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω και την κυρία Ζαπόρσκα για την εργασία της για το θέμα αυτό. Τρία θέματα που θα θέλαμε να τονίσουμε εγώ και οι συναδέλφοι μου στο στις τροπολογίες μας. Έχουμε την αίσθηση ότι ξαναξεκινάμε, γιατί όταν ε, ξεκίνησα τη δουλειά μου, έπαιρνα 15 ευρώ την εβδομάδα, ενώ οι άνδρες ε, συνάδελφοι έπαιρναν πολύ πιο πολλά. Και αυτό ήταν το 68 και σκεφτόμουν ότι δεν είναι δίκαιο και ακόμα το συζητάμε το θέμα αυτό. Συνεχίζεται. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν ποιες είναι οι συγκεκριμένες προτάσεις που μπορούμε να κάνουμε για να έχουμε αποτελέσματα. Δεν ε, μπορούμε να περιοριστούμε στο ότι α, παραπονιόμαστε, δεν είναι δίκαιο, να είμαστε επικοδομητικοί. Και αυτό θα ήθελα να κάνω με τις τροπολογίες μας. Καταρχάς, ο ρόλος των εθνικών σωμάτων ισότητας. Τα σώματα ισότητας θα πρέπει να έχουν αρμοδιότητες ε, ίσης μεταχείρισης ε, γυναικών και ανδρών σε θέματα απασχόλησης. Και αυτό ορίζεται σε αυτή την αναθεωρημένη οδηγία. Πολύ σημαντικό. Επίσης, ε, υπάρχει μεγάλη απόκληση στο, μεταξύ των κρατών ε, μελών. Σε κάποιες περιπτώσεις, το όνομα Βασίλειο στη Σουηδία έχει αρμοδιότητες στο σώμα αυτό. Σε άλλες περιπτώσεις, όπως η Γερμανία και στην Ιταλία, είναι λιγότερο αποδοτικά. Θα πρέπει λοιπόν να έχουν τις αρμοδιότητες, τους πόρους, το προσωπικό με τη σωστή εκπαίδευση, προκειμένου να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους και να μπορέσουν να λειτουργούν με τρόπο που θα εγγυάται την ανεξαρτησία τους από τις κυβερνήσεις. Όταν λειτουργούν με τον σωστό τρόπο, τα σώματα ισότητας μπορεί να έχουν σημαντική ε, επίδραση στην εφαρμογή της νομοθεσίας των κρατών μελών. Κατά δεύτερον, υποχρεωτικές, ε, υποχρεωτική έλεγχη με αμοιβή στις εταιρείες, στις μεγάλες εταιρείες. Θα αντισταθούν σίγουρα οι εταιρείες, αλλά υπάρχουν ε, μεγάλες διαφορές στην ε, αμοιβή. Με την εξαίρεση των μικρομεσαίων, εμείς προτείνουμε να υπόκεινται σε υποχρεωτικούς ελέγχους επί αμοιβής και έχουμε τεκμήρια από το Ενωμένο Βασίλειο που καταδεικνύουν ότι οι θελούσιοι έλεγχοι δεν έχουν τέτοια αποτέλεσμα. Στη τελική ανάλυση μόνο πέντε εταιρείε έκαναν αυτόν τον έλεγχο στο Ενωμένο Βασίλειο παρά το γεγονός ότι ήταν σχεδόν 300 αυτές που είχαν δηλώσει ενδιαφέρον ύστερα σε κάποια κρατημέλη σε ό,τι αφορά ότι τα προγράμματα εξειδότησης πρώτου, δεύτερου και τρίτου πυλώνα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις γυναίκες και στην πρόσβασή τους. Θέματα όπως το ωράριο, το μισθολογικό χάσμα, όλα αυτά επηρεάζουν το χάσμα στις συντάξεις. Και όλοι εξετάσουμε τα θέματα που απασχολούν τη σύνταξή μας και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει και τον αντίκτυπο στο χάσμα το συνταξιωτικό. Τέλος, ε, πρακτικές ε, που προστατεύουν τους πιο ευάλωτους. Ε, παρενόχληση, σεξουαλική παρενόχληση. Θα πρέπει να υπάρχουν καλοί κανόνες που θα έχουν βάση σε νομοθεσία, σε επίπεδο κρατικό αυτό μειώνει τις παρενοχλήσεις, γιατί ξέρουμε ότι όταν οι γυναίκες παρενοχλούνται έχουν την τάση να κάνουν πίσω. Δεν θέλουν απαραίτητα να πολεμήσουν. Αν υπάρχει μία δομημένη διαδικασία αναφορά τη παρενόχληση. νομίζω ότι αυτό θα τι βοηθήσει να αντιδράσουν καλύτερα. Αυτά θα βάλουμε λοιπόν στι τροπολογίε μα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Λόγοι Πρόεδρο, και τώρα το δίνω λόγο στην κυρία Ούμπερ. Ζούμπερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, να πω ότι αυτό που εμείς αντιλαμβανόμαστε για το όλο θέμα είναι το εξής. Η οδηγία όντως πρέπει να διατυπωθεί. Είναι πολλά τα νομοθετικά ζητήματα σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση και 100 μελών που μπορούν να βελτιωθούν. Να βελτιωθεί η ισότητα στον χώρο εργασία, αλλά ήδη υπάρχουν νόμοι, κάποιε φορέ είναι και καλοί, κάποιε φορέ προστατεύουν τι γυναίκε. Οπότε το βασικό ζήτημα είναι η σωστή υλοποίηση. Εδώ η Επιτροπή μα, από τη δική μα τουλάχιστον τη Σκοπιά, θα πρέπει να κάνει δουλειά, ε, μια σημαντική δουλειά, και να καταφέρει να ε, δείξει, να τονίσει ότι πολλές φορές η έλλειψη σωστής υλοποίησης της μεταφορά της νομοθεσίας για την ισότητα καλλιεργείται και από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την Τρόικα για διαφορετικούς λόγους. Εδώ υπάρχει μια σοβαρότατη αντίφαση μεταξύ της νομοθεσίας και μεταξύ των όσων είναι μακροοικονομικές πολιτικές και ο συντονισμός τους ε, ή ε, τα ευρωπαϊκά όργανα επιβάλλουν στα κράτη-μέλη. Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε αυτό το στοιχείο που φαίνεται να είναι σε ένα βαθμό προφανές. Πρέπει λοιπόν με τις τροπολογίες που έχουν προταθεί να βελτιώσουμε την έκθεση γιατί συμφωνούμε με την ε, φιλοσοφία της έκθεσης την, τα όσα έχει συμπεριλάβει η συνάδελφος Ζαμπόρσκα, αλλά πρέπει να προσδέξουμε και τα εξή. Τι ισχύει με τις συλλογικές συμβάσεις. Εδώ θεωρούμε ότι οι ποσοστώσεις φαίνονται και από την πολύ σκληρή ε, Μάλλον οι ποσοστώσεις επηρεάζουν και, επηρεάζονται και από τη σκληρότατη τη φορολογία. Δούμε τα με, τη μελέτη για την ανάπτυξη του 2015. Βλέπουμε ότι τα κράτη-μέλη στρέφονται κατά των συλλογικών συμβάσεων και ε, για, ότι η συλλογική δράση τελικά δεν ε, ε, επιτρέπεται με τα νέα μέτρα των κρατών μελών. Εδώ πλήττεται και η ισότητα. Και αυτό πρέπει να τονίσουμε. Πρέπει λοιπόν να δούμε τον εργασιακό χώρο ε, από τη σκοπιά της μισθολογικής και της αυτοαξιολόγησης των εργαζομένων και αυτό μας φαίνεται εξαιρετικά σημαντικό και προφανώς ό,τι έχει να κάνει με το με την ε, φορολόγηση και την ε, εφαρμογή του νόμου από το κράτος τους και τους κρατικούς φορείς. Εδώ αν δεν δούμε την πραγματικότητα κατάματα, εάν ε, δεν εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη στους κρατικούς φορείς τους κανόνες του εργατικού δικαίου, τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την εργασία, Όλα αυτά δεν θα καταφέρουν ποτέ να υλοποιηθούν σωστά. Υπάρχει λοιπόν μια κατάσταση πολύ ευάλωτη. Ε, η ανεργία αυξάνεται. Δεν θα αλλάξει η πραγματικότητα, διότι όλοι γνωρίζουμε ότι η ανεργία φέρνει τους εργαζόμενους ακόμη πιο επισφαλή θέση. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι γίνεται στον εργασιακό χώρο ε, και όχι μόνο μία φορά, δύο, τρεις και τέσσερις για να μπορέσουν να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη τους οι εργαζόμενοι και να ε, ξέρουν ότι προστατεύονται. Ε, όταν κανείς θεωρητικά καταλαβαίνει και αντιλαμβάνεται τον νόμο, ακόμα και να διακριτική μεταχείριση στις γυναίκες σε εταιρείε ή εργοστάσια, θα πρέπει να δούμε γιατί οι γυναίκες πηγαίνουν στις χαμηλότερες ε, επαγγελματικέ κατηγορίες, εκεί που αδιακρίτως δουλεύουν οι εργαζόμενοι. Το πρόβλημα λοιπόν είναι η θέση εργασία. Είναι, όταν μιλάμε με τι γυναίκε επί τη ουσία, βλέπουμε ότι του ζητάτε μια ευελιξία για να μπορέσουν να καλύψουν επαγγελματικά καθήκοντα που αντιστοιχούν σε άλλα προσόντα και που πολλέ φορέ τα καλύπτουν κανονικά άντρε. Πρέπει λοιπόν να δούμε ε, την πραγματικότητα συζητώντα με τι επιχειρήσει και τι εταιρείε οι εταιρείε πρέπει να ευαισθητοποιηθούν για το θέμα. Διότι αν ε, καταλάβουν ότι του φέρνει μεγαλύτερο κέρδο το να λάβουν υπόψη του αυτή τη διάσταση, θα το κάνουν. Το θέμα είναι να ε, είμαστε λοιπόν ε, πραγματιστές στην προσέγγιση μα και να επιβληθούν και πρόστιμα κυρώσει. Διότι δεν υπάρχει λόγο να πληρωθεί απλώ ένα πρόστιμο σε περίπτωση παραβιάζει των νόμων. Δεν αρκεί αυτό. Διότι αν μπορεί με ένα μια επιχείρηση να παραβαίνει τον νόμο, θα συνεχίσει να το κάνει. Ε, υπάρχουν και άλλε τροπολογίε που επιβάλαμε, που έχουν να κάνουν με άλλε λεπτομέρειε. Θεωρούμε όμω ότι οι εργαζόμενε βρίσκονται σε θέση ευάλωτη σε σχέση με τον εργοδότη, με το αφεντικό. Θα πρέπει λοιπόν οι εταιρείε να καταγγείλουν, οι εταιρείε να προβλέψουν τα απαραίτητα μέτρα, να αποδείξουν ότι δεν παραβιάζουν τον νόμο, ότι δεν ασκούν διακριτική μεταχείριση. Εν τέλει, να πω στη συνάδελφο Ζαμπόρσκα, όπου μιλάει για συμφιλίους οικογενειακού και επαγγελματικού βίου, και λέει ότι μια από τι καινοτομίε, τι οδηγίε κλπ. κλπ. Εδώ βρίσκω ότι υπάρχει και άλλη αντίφαση τη ίδια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι αυτό που βλέπουμε είναι να αυξάνονται τα ωράρια εργασία ε, και ζητάτε μεγαλύτερη ευελιξία ω προ το ωράριο εργασία από του εργαζομένου. Αυτό δεν συνάδει με τη συμφιλίωση οικογενειακού επαγγελματικού βίου, κάτι πρέπει να διαλέξουμε. Είναι σαφέ. Δεν μπορούμε να εφαρμόζουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δεν μπορούμε να ζητάμε ένα πράγμα και το αντίθετό του ταυτόχρονα. Πρέπει να γίνουν επιλογέ και να καταγγελθούν ε, οι υπεύθυνοι για να αναλάβουν και τι ευθύνε του. Από πολιτική τουλάχιστον σκοπιά. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Η ε, κυρία το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ την συνάδελφο την Άννα Ζαβρόφσκα και συγχαρητήρια. Ακόμα για να έχουμε 169 τροπολογίες, δύσκολα θα πρόσθετα κάτι γιατί είναι αρκετά πλήρης και αρκετά σύνθετη η έκθεσή σας, το κείμενό σας, αλλά μία τροπολογία θα μπορούσα να προσθέσω για να υπογραμμίσω το βασικό πρόβλημα για τις γυναίκες. Όταν γυρνάνε στη δουλειά, η δυσκολία που έχουν να ξαναβρούνε το μισθό τους, η σταδιοδρομία τους επαγγελματική είναι πάντα πιο περιορισμένη. Περιορίζεται από το φυσικό τους ρόλο που είναι η μητρότητα. Πάντα συμβαίνει αυτό. Αν λοιπόν θέλουμε να κάνουμε κάτι για να υπάρχει ισότητα αμοιβών και συνθήκων, πρέπει να βελτιώσουμε τις συνθήκες για τις γυναίκες. Όταν επιστρέφουν στη δουλειά μετά τη μητρότητα, αλλά και ώστε να δίνουμε την αξία που πρέπει στη μητρότητα. Αυτό είναι κάτι που θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, ευχαριστώ. Πριν δώσουμε το λόγο στην κυρία Ζαμπρόφσκα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλω να ρωτήσω. Μήπως έχει κάποιον εδώ που θέλει το λόγο. Όχι. Ωραία, κύριε Ζαμπρόσκα τότε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις ε, από τους συναδέλφους, από τις συναδέλφους. Σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Είναι πολύ ενδιαφέρον να ακούμε αυτά που είπατε. Αν από πλευρά της ε, κοινωνίας δεν ε, γινόντουσαν προσπάθειες να αλλάξει η κατάσταση, τι να μας βοηθούσαν δέκανες ε, οδηγίες. Άχρηστες θα ήτανε. Πάντα θα ήμασταν αντιμέτωπες τελικά με την ίδια κατάσταση. Και γι' αυτό λοιπόν θέλω να ζητήσω το εξής. Ένα από τα επόμενα έτη να αφιερωθεί στην ισότητα τη μισθολογική μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να ευαισθητοποιηθεί στο πρόβλημα αυτό που υπάρχει. Είμαι απόλυτα πεπισμένη ότι πολλοί δεν το γνωρίζουν καν το πρόβλημα. Είναι όμως πολύ σημαντικό και για την καλύτερη εκπαίδευση των γενικών. Θα πρέπει και αυτό να το φροντίσουμε σε κάθε περίπτωση. Και θα πρέπει να αντιληφθούμε το εξής. Ότι θα πρέπει να υπάρχει ίσια εργασία σε ίσο επίπεδο εκπαίδευσης. Αυτό τι σημαίνει. Ότι ίσως οι καλύτερα εκπαιδευμένες γυναίκες θα πρέπει να έχουν καλύτερες θέσεις. Το θέμα όμως της διαφοράς του μισθού δεν επιλύεται και πάλι με τον τρόπο αυτό. Φυσικά όμως θα πρέπει να φροντίσουμε να είναι καλύτερη εκπαίδευση των γυναικών. Αντελή έκανε στο σημείο αυτό μια σημαντική παρατήρηση. Ότι η δουλειά των γυναικών ως μητέρες δεν συνυπολογίζεται στο καθάριστο εθνικό προϊόν. Και αυτό δημιουργεί διαφορές και ανισότητες στους μισθούς. Ανέφερα και την πρώτη προηγούμενη φορά ότι το θέμα της μισθού και της μισθολογικής ε, διαφοράς εντοπίζεται μετά την επιστροφή της γυναίκας ε, στην, ε, στο χώρο εργασίας μετά την πρώτη γέννα. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν σχετικές κυρώσεις. Έγινε μια εντατική συζήτηση σχετικά με αυτό ήδη το έτος 2006 με την έκθεση της Edith Bauer για το μισθολογικό χάσμα. Θα ήθελα να καλέσω λοιπόν τους συναδέλφους ε, να συνειδητοποιήσουν ότι θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές ό,τι αφορά τις κυρώσεις. Σήμερα έχουμε ένα ψήφισμα, ψηφίσαμε ένα ψήφισμα για τη μητρική άδεια. Αυτό ήταν απαραίτητο λοιπόν. Πριν από 5-6 χρόνια το Κοινοβούλιο είχε δείξει υπερβολικό βαθμό φιλοδοξίας. Αυτό τι σημαίνει. Αν θέλουμε να πετύχουμε αλλαγέ στην οδηγία, θα πρέπει να υπολογίσουμε και το Συμβούλιο και το ρόλο του Συμβουλίου. Γιατί αν θέσουμε υπερβολικά μη ρεαλιστικές ε, προσδοκίες, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου τελικά δεν εκπληρώνεται κανένα όνειρο των γυναίκων. Δεν βελτιώνεται σε τίποτα η θέση των γυναίκων. Υπολογίζω λοιπόν στην βοήθειά σας προκειμένου για να θεώρηση αυτή να ψηφιστεί στην Ολομέλεια με την μεγαλύτερη δυνατόν πλειοψηφία. Ελπίζω και βλέπω ότι υπάρχει αυτή η ελπίδα γενικότερα Είμαι ανοιχτή φυσικά σε τροπολογίες ε, που θα καταθέσετε. Αλλά θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και ρεαλίστρες για να πετύχουμε μια ενιαία άποψη και μια ενιαία τοποθέτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα πρέπει το κείμενο να γίνει αποδεκτό και από το Συμβουλίο. Τέλος. Ευχαριστώ όλους και όλες για τις προτάσεις ε, τροπολογιών. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Ήταν ε, το τελευταίο αυτό σημείο αυτό στην ημερήσια διάταξη. Η ψηφοφορία θα γίνει 15 και 16 Ιουνίου, όπως αναφέραμε ήδη. Έχουμε πολλές καλές συναντήσεις μέχρι τότε, προκειμένου να πετύχει η έκθεση. Αύριο θα τα πούμε στις 9 ώρες. ευχαριστώ πολύ.